Good uh, Καλώς λοιπόν, περιμέναμε 10 λεπτά για τους συναδέλφους. Ελπίζω να εμφανιστούν οι υπόλοιποι. Σας καλωσορίζω λοιπόν όσοι είστε εδώ. Ευχαριστώ που ήρθατε εγκαίρως. Θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. έχουμε μια πρόταση γνωμοδότησης με την κυρία Τζουφρίντα. Ετήσια έκθεση 2015 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πολέμηση των απατών. Το άρθρο 220, σύμφωνα με το άρθρο 225 δημοσιεύει μια έκθεση η Κομισιόν για τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση της απάτης. Καλύπτουμε όλους τους τομείς. Η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού κάνει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας πάνω στην έκθεση της Επιτροπής για το 2015 και η δική μας Επιτροπή συντάσσει μια γνωμοδότηση. Η κυρία Τζουφρίντα θα παρουσιάσει την πρότασή της Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 12 το μεσημέρι. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Τζουφρίντα και μετά στους Κιώδης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινώντας να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ετήσια έκθεση για το 2015 που μας έδωσε σημαντικά στοιχεία περιληπτικά λέγεται ότι το 2015 παραπέμφθησαν στα κράτη-μέλη 23.349 μη κανονικές ε, δαπάνες. Από αυτές 1.461 σημειώθηκαν ως απάτες. Τα υπόλοιπα είναι απλά ε, έλλειψη τακτικής δημοσιονομικής πρακτικής. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να εμβαθύνουμε στο φαινόμενο της απάτης. Νομίζω ότι απαιτείται μια πραγματικά μεγαλύτερη προσοχή έτσι ώστε να δούμε αν τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας είναι κατάλληλα για την αξιολόγηση των απατών. Γι' αυτό ακριβώς έπρεπε να συλλέξουμε τις περισσότερες τεκμηριώσεις στις 10 Οκτωβρίου συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της Όλαφ και της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζο. Φιλοξενήσαμε και τον Γενικό Διευθυντή και τους εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη που είναι υπεύθυνοι για τις απάτες. Είδαμε ποια είναι τα προβλήματα που επέτρεψαν να γίνουν οι απάτες αυτές και πώς όταν γνωστοποιηθούν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν το σύστημα. Πάρα πολύ συχνά η συγκέντρωση συγκεντρώνεται στην δυνατότητα χρήσης των πιστώσεων αυτών από τις ε, τοπικές αρχές και τις εθνικές αρχές. Η ποιότητα όμως ε, του τρόπου με τον οποίο θα πανώνται οι πιστώσεις αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε λοιπόν ότι η ιστορία με τις απάτες δεν είναι μια προσπάθεια για να ανακτήσουμε μια μικρή οικονομική βλάβη αλλά είναι αναπόσπαστο τμήμα και χαρακτηριστικό της πολιτικής μας στον τομέα. Νομίζω ότι δεν εμβαθύνει πολύ στην πολιτική συνοχή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά οι έρευνες που έγιναν το 2015 νομίζω ότι μας δείχνουν ακριβώς σε ποια επίπεδα πληρωμών φτάσαμε. Γίνονται βέβαια προσπάθειες για να εμβαθύνουμε τον συσχετισμό ανάμεσα στις απάτες από τη μία και τα τα μία από την άλλη. Η Όλαφ έχει μια από την άλλη. Η Όλαφ έχει μια ειδική ερευνητική ομάδα για τα διαφθορτικά. Να δούμε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Όπως έλεγα, οι απάτες που ανακοινώθηκαν από τα κράτη-μέλη είναι πάνω από 22.000. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια αξιολόγηση ε, ε, μιας, ε, ενός καταλόγου θα έλεγα, ο οποίος να δείχνει σε ποιες χώρες γίνονται πολλές απάτες και σε ποιες όχι. Πραγματικό... Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, αλλά είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών να προστατεύουν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που άπτεται και της προστασίας των εθνικών οικονομικών συμφερόντων. Γι' αυτό λοιπόν ο τρόπος και ο τακτικός ημί, ο τακτός μάλλον η μη χαρακτήρας των αναφορών των κρατών μελών είναι κάτι το οποίο γίνεται με τρόπους που επιλέγουν τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να μπορέσουμε βέβαια να κάνουμε συγκρούσεις, αλλά οι αριθμοί από μόνοι τους δεν μας λέγουν το τι συμβαίνει. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια περαιτέρω ομογενοποίηση των στοιχείων αυτών. Η συλλογή των περιπτώσεων απανών που θα χρησιμοποιηθεί για να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στις εισαγωγικά διεφθαρμένες χώρες και στις χώρες χωρίς απάτες είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Ε, στο αρχείο πηγαίνουν οι, περισ... οι λιγότερες από τις καταγγελίες και η έλλειψη αυτή του σεβασμού των κανόνων οφείλεται στις δυσκολίες πολλές φορές των διαδικασιών. Γι' αυτό ακριβώς από τη μία αναφερόμαστε στην ανάγκη εντατικοποίησης της τεχνικής αρρωγής των δημοσίων διοικήσεων και από την άλλη την απόλυτη αναγκαιότητα να υπάρξει μια περαιτέρω απλούστευση της πολιτικής συνοχής. Υπό το φως λοιπόν αυτών τα οποία είπα και βλέποντας πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα και πόσο σχετικά είναι τα δεδομένα, τίθεται εδώ το θέμα της αξιοπιστίας της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να προσέξουμε τη χρήση των στοιχείων αυτών και να επιτρέψουμε στην Ευρώπη σε μια μάλιστα δύσκολη περίοδο να προχωρήσει. Οι απάτες στην πολιτική συνοχή είναι σοβαρές και είναι σοβαρές διότι βλάπτουν το σύνολο των πολιτών. Αλλά ευτυχώς μέχρι τώρα φαίνεται να ανοιχνεύονται από τις αρχές των κρατών μελών και της Ένωσης και δεν είναι σε ιδιαίτερα μαζικό επίπεδο. Πρόκειται για έρευνες οι οποίες ολοκληρώνονται πολλές φορές χωρίς αποτελέσματα και ενώ ε, κάποια ποσά ανακτώνται, άλλοτε προβλέπονται άλλοι μηχανισμοί διαχείρισης. Αν θέλουμε εμείς να καταστήσουμε τα συστήματα πιο αξιόπιστα, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην πρόληψη και όχι μόνο στην καταστολή Γι' αυτό ακριβώς η διοικητική συνδρομή είναι χρήσιμη. Πρέπει να υπάρξει και μια καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις διαχειριστικές αρχές και στις αστυνομικές αρχές μέσω μνημονίων κατανόησης που διαθέτουν τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στις δύο πλευρές. Τα όρια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν τεθεί δεν επιτρέπουν να τα ποσοτικά όρια, να σας δώσω περισσότερα στοιχεία, αλλά θα προσπαθήσω να ενσωματώσω τις προτάσεις όλων των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους κοιότητες εισηγητές, ξεκινώντας από τον κύριο Γιάκο Φτσίτς. Θα μας παρουσιάσει την άποψη της κυρίας Νικολάη. Καλά το είπα, Μα, μάλιστα. Μις Νικολάη, Νικολάη, Ναι, θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να, εξασφαλίσουν ότι και οι, προστα... και οι φορολογούμενοι και ο προϋπορισμός τη Ένωση την χάνει τη απαιτούμενη προστασία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση ότι τα κονδύλια δαπανούνται για του στόχου τους, ε, ε, για του οποίου διατέθηκαν και θα ωφελούν του πραγματικού ε, δικαιούχου. Οι εθνικέ αρχέ θα πρέπει να μπορούν να επαληθεύουν τι χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι παρατηρούνται παρατυπίες είτε στις διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμών είτε σε άλλα επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προετοιμάσουν ένα σύστημα που θα βασίζεται στην πρόληψη, αλλά και να ενισχύσουν τις αρχές με ερευνητικές, ελεγκτικές εξουσίες για να προστατευτούν τα χρηματοπιστωτικά συμφέροντα της Ένωσης. Η ε, Όλαφ είναι ένα σημαντικό θεσμός θα πρέπει να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει όμως επαρκή επικοινωνία. Αυτό πρέπει να βελτιωθεί αν θέλουμε να μειωθεί η απάτη και να ανακτηθούν τα κονδύλια. Γιατί πέραν της βελτιώσης της επικοινωνίας μεταξύ όλων και κρατών μελών, υπάρχει ανάγκη ευαισθητοποίησης ε, και ενημέρωσης και των Ευρωπαίων πολιτών για την αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης της απάτης τα οποία έχουν εγκριθεί Επίσης πρέπει να αυξηθεί διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης ε, των σχεδίων τα οποία υλοποιούνται με εξωτερικά κονδύλια. Τέλος, για να εξασφαλιστεί η προστασία των χρηματοπιστωτικών σφαιρόντων της Ένωσης, η πρόταση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου, του Γραφείου Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα είναι κάτι θετικό για ενίσχυση των μέτρων της καταπολέμησης και πρόληψης της απάτης. Αυτά τα είπε η συνάδελφος Νικολάη. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. νταμάτο, κυρία, εσείς είστε συγγήτρια επίσης, σκιώδης. Ευχαριστώ τη συνάδελφο για τη δουλειά την οποία έκανε. Η έκθεσή της είναι σημαντική για την προστασία των συμφερόντων των οικονομικών της Ένωσης. Κάποια επιπλέον στοιχεία Συμφωνώ σαν παράδειγμα για την ανάγκη μιας πραγματικής εναρμόνισης της ταξινόμησης των συμβάντων και της αναφοράς των συμβάντων. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην οφειλόμενη διοικητική επιφυλακτικότητα, η προσοχή αν θέλετε, και από την άλλη στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Ένα ειδικό θέμα είναι οι προμήθειες, οι διαγωνισμοί για προμήθειες, Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να υπακούσουμε στις συστάσεις του ε, Συμβουλίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου μάλλον, η πολιτική σύνοχης ε, δεν ήταν η πολιτική με τις περισσότερες μη τακτές ε, οικονομικές ενέργειες. Παρόλα αυτά το ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύει οικονομικά είναι υψηλό. Υπάρχουν επίσης ε, πάρα πολλές ε, παραβάσεις ε, των κανόνων των δημοσιονομικών, γι' αυτό θα πρέπει η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές να συνεχίσουν την προσπάθεια καταπολέμησης των απατών για να μην θίξουμε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής που είναι κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη αλλά είναι πολύ περιπλοκή και δεν γίνεται κατανοητή από τους συμπολίτες μας. Thank you. Are there... Ευχαριστώ. Άλλος κανείς. Κύριε Μπρέσο, ναι, γνωρίζω. Εκπροσωπείτε τον σκιώδη συγκητή, τον κύριο Ρόπιν, την κυρία Ρέγκη. Εντάξει, πρώτα εσείς κύριε Μπρέσο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την συνάδελφο για μια συγκεκριμένη έκθεση, μια έκθεση γεμάτη από προτάσεις χρήσιμες. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το σύνολο της πολιτικής σύνοχης. Οι επιθέσεις πολλές φορές εναντίον της πολιτικής σύνοχης βασίζονται στον αριθμό των απατών ή μη τακτικών οικονομικών ενεργειών και λαμβάνουν υπόψη αυτά τα οποία είπε η συνάδελφος, λαμβάνουν υπόψη τους αριθμούς οι οποίοι δεν είναι επιβεβαιωμένοι βέβαια, αλλά αποτελούν αντικείμενο καταγγελίας. Συνεπώς λοιπόν, από τη μία, ένα μεγάλο τμήμα των περιπτώσεων αυτών οφείλεται, όπως είπε η συγγήτρια, στον περίπλοκο χαρακτήρα των διαδικασιών. Οπότε είναι πολύ λογικό να υπάρξουν λάθη, να υπάρξουν ε, ε, πραγματικά κάποιες προσπάθειες ερασιτεχνικές απλοποίησεις, αλλά και η προσπάθεια της Επιτροπής στον τομέα της απλοποίησης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς η σχέση ανάμεσα, πώς φαίνεται να αναπτύσσεται η σχέση ανάμεσα στην απλούστευση από τη μία και στις μη τακτές ε, ε, οικονομικές ε, ενέργειες από την άλλη μπορούμε να κάνουμε ένα συσχετισμό για να δούμε ακριβώς τι χρειάζεται στον τομέα της υπεραπλούστευσης, να μην φτάσουμε μάλλον στην υπεραπλούστευση. Αν εμείς πράγματι θέλουμε να υπάρξει μία σύγκριση φέρνοντας εδώ στις Βρυξέλλες, όπως το πρότεινε και η συνάδελφος, τους υπευθύνους των διαχειριστικών αρχών των εθνικών που εμπλέκονται στις διαδικασίες αυτές για να καταλάβουμε με συγκεκριμένο τρόπο πώς μπορούμε εμείς να απλουστεύσουμε τα πράγματα έτσι ώστε να μειώσουμε ε, αυτές τις απάτες ε, και τις μη τακτικές οικονομικές ενέργειες. Υπάρχουν και απάτες ε, <clears throat> και εάν καταφέρουμε να μειώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο μέσω της απλοποίησης, αυτό θα είναι μια προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ. Τώρα, κύριε Ροπέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό οι λύσεις που θα προτείνουμε θα είναι αποφασιστικές για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να σκεφτούμε την παρούσα προγραμματική περίοδο καθώς και το διάστημα μετά το 2020. Έχω κάποιες παρατηρήσεις και κάποιες ερωτήσεις, διότι με ανησυχεί η κατάσταση. Σε ποια κράτη-μέλη βλέπουμε τις περισσότερες παρατυπίες. Ε, μπορεί να μην χρειαζόμαστε τον ε, αριθμό των παρατυπιών, αλλά ε, τα χρηματικά ποσά που αφορούν. Και τι οδηγεί στις παρατυπίες αυτές. Επίσης, μπορούμε να τις συνδέσουμε με απάτες που συνδέονται με εθνικούς πόρους. Εάν δηλαδή το είδος της απάτης είναι παρόμοιο και όταν μιλάμε για τον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και για τον εθνικό, τότε το πιθανότερο είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν κακό σύστημα διοίκηση και ότι χρειάζονται τη βοήθειά μας για να βελτιώσουν το σύστημα ε, δημοσιονομικής διαχείρισης. Όσον αφορά τις απάτες, είναι σημαντικό να μιλάμε για την αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων, διότι η μη αποτελεσματική απορρόφηση έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την απάτη. Εάν δεν δαπανούμε ε, ε, αποτελεσματικά, με αποτελεσματικό τρόπο τα χρήματα, τότε ε, αυτό δεν ωφελεί ούτε την Ευρώπη, ούτε τα κράτη-μέλη, ούτε τους πολίτες. Επί δέκα χρόνια ήμουν αρμόδιος για την δαπάνη ευρωπαϊκών πόρων σε μια τοπική αρχή. Πολλοί θεωρούν το ευρωπαϊκό χρήμα δώρο. Δεν θεωρούν ότι είναι χρήματα των φορολογουμένων πολιτών. Και νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στους απλούς ανθρώπους ώστε να καταλάβουν ότι και, το, και οι ευρωπαϊκή πόροι είναι ε, χρήματα που προέρχονται από τους φορολογούμενους ε, και εάν ε, κάνουν απάτες που έχουν να κάνουν με αυτούς τους πόρους, τότε κλέβουν τον φορολογούμενο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μια περιφέρεια όπου μια τοπική περιφέρεια ε, καταφέρνει να εξοικονομήσει κάποια χρήματα. Αλλά ε, τα χρήματα αυτά που εξοικονομεί δεν παραμένουν εκεί. Ε, τα παίρνουν πίσω. Για παράδειγμα, κατασκευάζεται ένας δρόμος με 100 εκατομμύρια ευρώ. Ε, για ένα εκατομμύριο ευρώ. 900.000 ε, μπορεί να προσφέρει ένα ε, εργολάβο, αλλά δεν έχουν κίνητρο να εξοικονομήσουν αυτές τις 100.000, διότι θα σταλούν πίσω στην κεντρική αρχή και έτσι θα χάσουν τα χρήματα αυτά. Έτσι προτιμούν να δαπανίσουν ολόκληρο το εκατομμύριο. Ενώ εάν είχαν τη δυνατότητα να κρατήσουν τα χρήματα που έχουν εξοικονομήσει, θα είχαν περισσότερα κίνητρα. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η αποκέντρωση. Κατά τη γνώμη μου, εάν καταφέρουμε να έχουμε κεντρική διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, η επιρροή πολιτικών κομμάτων και πολιτικών ε, γενικά θα είναι σημαντική. Αν καταφέρουμε να αποκεντρώσουμε την ε, δαπάνη και να δώσουμε περισσότερες ε, ευθύνες σε τοπικό επίπεδο, πιστεύω ότι θα μειωθούν οι παρατυπίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τους ευρωβουλευτές. Ε. Α, ο κύριος Νοβάκοφ, παρακαλώ. Υποθέτω ότι ήρθατε για να μιλήσετε για το θέμα αυτό. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Βούλα για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ως σκιώδης εισηγητής στην έκθεση αυτή. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά που συζητάμε αυτή τη στιγμή και έχουμε κακά νέα. έχουν αυξηθεί οι παρατυπίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά περισσότερο από 30%. Αυτό σίγουρα είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε. Ένας από τους λόγους που έχουμε περισσότερες ε, παρατυπίες αυτή τη στιγμή είναι οι πολύπλοκες νομοθετικές διαδικασίες. Ε, αυτή τη στιγμή λοιπόν μιλάμε για παρατυπίες, όχι για απάτη. Ποιες είναι οι πιθανές λύσεις η απλούστευση και χαίρομαι που αυτή αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή Ρέτζη. Δεύτερον, χρειαζόμαστε πιο στενή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να αποφεύγουμε τέτοιες πρακτικές που οδηγούν σε παρατυπίες. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει μια καλή αρχή. Θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους εταίρους μας για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση. Διότι δεν ε, αυξάνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών οι περισσότερες παρατυπίες. Ε, εφόσον λοιπόν έχουμε ένα σύστημα θα πρέπει ε, τους ευρωπαϊκούς σπόρους να τους ε, κατανείμουμε Ε, στους ε, διάφορους φορείς, αλλά το 30% των παρατυπιών που έχουμε δεν βοηθάει στο να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη ε, των ψηφοφόρων μας. Νομίζω γενικά ότι έχουμε πετύχει πολύ καλή ισορροπία στην έκθεση. Προσβλέπω στις επόμενες συζητήσεις πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε τον κύριο ε, Ανδρέα Μπορδόνη από την Όλα. Θα θέλατε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι ένας από τους βασικούς ε, συνσυντάκτες ε, της έκθεσης, ιδιαίτερα όσον αφορά το στατιστικό κομμάτι. Ελπίζω λοιπόν να μπορώ να σας δώσω κάποια στοιχεία για καλύτερη κατανόηση της στατιστικής πτυχής της έκθεσης αυτής ιδιαίτερα. Καταρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι η έκθεση αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για να καταπολεμήσουν την απάτη και τις παρατυπίες. Γι' αυτό έχουμε δύο πτυχές εδώ, την πολιτική πλευρά, όπου τονίζουμε τα πολιτικά μέτρα σε νομοθετικό ή διοικητικό επίπεδο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίπεδο κράτους μέλους ε, για να καταπολεμηθούν ε, οι παρατυπίες και οι απάτη και να προστατευτούν ε, τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, έχουμε τα αποτελέσματα των περιπτώσεων παρατυπίας ή απάτης που έχουν εντοπιστεί από τις εθνικές αρχές και που έχουν αναφερθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο Όλαφ που ε, διαχειρίζεται το σύστημα διαχείρισης των παρατυπιών το κάνει αυτό ε, στο όνομα υπηρεσιών της Επιτροπής. Λαμβάνουμε τις πληροφορίες αυτές, τις επεξεργαζόμαστε και ενημερώνουμε εσάς και το Συμβούλιο με την έκθεση αυτή. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο. Υπό το φως αυτό θα πρέπει να δείτε την έκθεση αυτή και τα δεδομένα που αναφέρουμε. Δεύτερη, δεύτερο, δεύτερη παρατήρηση είναι η συγκρισιμότητα των δεδομένων. Κάνουμε πολλή δουλειά πάνω στο θέμα αυτό. Όλο το φετινό έτος ε, το έχουμε αφοσιώσει στην ε, εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών από ε, εμπειρογνώμονες από 14 μέλη ε, για να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί κατά την εξέταση των παρατυπιών. Αύριο έχουμε άλλη μια συνάντηση με τους εθνικές, εθνικούς εμπειρογνώμονες και προσπαθούμε το τελικό αυτό έγγραφο για με τις κατευθυντικές γραμμές ε, και για την υποβολή των εκθέσεων να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος της χρονιάς ή μέσα στους πρώτους μήνες ε, του επόμενου έτους. Αυτός είναι ο στόχος μας. 1η ε, Απριλίου του 2016 κυκλοφόρησε η νέα εκδοχή του συστήματος διαχείρισης των παρατυπιών που ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές να έχουν καλύτερη πρόσβαση Προσπαθούμε λοιπόν να παράσχουμε επαρκή εργαλεία για την ε, υποβολή ε, εκθέσεων. Επίσης, ε, όσον αφορά την αύξηση ή πτώση των παρατυπιών που αναφέρονται, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πάντα πολύ δύσκολο να εντοπίσει κανείς τους, τις αιτίες, διότι οι παρατυπίες που φτάνουν σε εμά διαπιστώνονται περίπου τρία χρόνια μετά. Ε, το 2015 λοιπόν ε, μιλάμε για πράγματα που έχουν συμβεί το, 2015, ε, το 2012 κατά μέσο όρο και θα πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Δεύτερον, πάντα υπάρχουν πολλοί λόγοι αύξησης ή μείωσης που προσπαθούμε να εξηγήσουμε στην έκθεση. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά σαφείς. Ε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα πολιετή και τα μονοετή προγράμματα. Ε, στα πολιετή προγράμματα υπάρχει μια ε, φυσική τάση. Όσο λοιπόν εφαρμόζονται τα προγράμματα στα κράτη-μέλη, τόσο περισσότεροι πόροι διατίθενται, δαπανώνται και γι' αυτό έχουμε και περισσότερες παρατυπίες και γι' αυτό έχουμε αύξηση για μια σειρά ετών και μετά απότομη πτώση. Φέτος είχαμε μια ιδιαίτερη κατάσταση που αναφέρεται στην έκθεση που συνδέεται με την πολιτικη συνοχή. συνοχής. Έχουμε δύο κράτη-μέλη, την Ισπανία και την Ιρλανδία, που ανέφεραν ε, μεγάλο όγκο παρατυπιών πολλά χρόνια ε, αφότου θα έπρεπε να το έχουν κάνει. Ε, αυτό λοιπόν αλλάζει κάπως την εικόνα. Το 36% των παρατυπιών που αναφέρονται για το Ταμείο Συνοχής το 2015 είναι τέτοιες περιπτώσεις. Τέλος, ε, για να μην μακρηγορήσω και να μην σας φορτώσω με υπερβολικά πολλές ε, πληροφορίες, όσον αφορά τις ε, παρατυπίες που αναφέρονται ως δόλιες, εδώ μιλάμε για ανάλυση της προοπτικής για τα τελευταία χρόνια. Η διαπίστωση απάτης δεν είναι πάντα εύκολη. Πάντα ε, αναφέρουμε ένα στοιχείο της απάτης που είναι η πρόθεση. Το δεύτερο στοιχείο όμως είναι η απάτη. Κάποιος λοιπόν που προσπαθεί να εξαπατήσει ένα θύμα μέσω του κυβερνοεγκλήματος, ε, μέσω κανονικής απάτης ή στα διαφορετικά ταμεία, υποβάλλει ε, έγγραφα με ψευδή στοιχεία. Για να διαπιστώσουμε λοιπόν ότι τα στοιχεία αυτά είναι ψευδή, χρειάζεται να γίνουν εις βάθος έρευνες. Μπορεί λοιπόν τα έγγραφα που έχετε λάβει να φαίνονται απόλυτο σωστά, μόνο όμως ε, αφού ε, αφού διεξάγουμε διασταυρούμενους έλεγχους και μάλιστα συχνά με φορείς που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος από ότι το κράτος μέλος από το οποίο προέρχονται τα έγγραφα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι πράγματι έχει υπάρξει απάτη. Όποτε λοιπόν έχουμε περιπτώσεις πιθανής απάτης που υποβάλλονται σε εμά, ε, έχουμε τέτοιες ε, εις βάθος έρευνες. Και Γι' αυτό λέμε ότι ε, έχουμε ενδείξει ότι αυτό το σύστημα κατά της απάτης ε, λειτουργεί. Και γι' αυτό μπορούμε επίσης να πούμε ότι είναι πολύ μικρός αριθμός των ε, δόλειων παρατυπιών σε σχέση με τα χρήματα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Εάν όμως ε, έχουμε να πούμε κάτι για τα κράτη-μέλη Οι περιπτώσεις όπου δεν αναφέρονται ε, περιπτώσεις παρατυπίας για πολλά έτη το ένα μετά το άλλο. Ε, αυτό θα το δείτε στο σημείο 3 της έκθεσης. Σε μία τελευταία παρατήρηση για την απλούστευση. Νομίζω ότι θα πρέπει να δεχτούμε ένα στοιχείο. Η πολιτική συνοχής είναι ένα πολύπλοκο πλαίσιο. Μιλάμε για πολλές, πολλά επίπεδα αρχών πολλά επίπεδα νομοθεσίας. Ε, για παράδειγμα, έχουμε την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις που πρέπει να μεταφερθεί σε εθνικό επίπεδο. Κατόπιν ε, έχουμε το περιφερειακό επίπεδο για τα προγράμματα. Ε, μετά μπορεί να έχουμε έναν Δήμο που λαμβάνει χρήματα για ένα πρόγραμμα και ξεκινάει τη δική του διαδικασία Δημόσια σύμβάση. Ε, και σε όλα αυτά τα επίπεδα μπορούν να εφαρμοστούν με διαφορετικό τρόπο οι κανόνες. Πρέπει να δεχτούμε ότι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το σύστημα. Έχει ε, επιλεγεί η αποκεντρωμένη προσέγγιση, επειδή έτσι προσεγγίζουμε καλύτερα τους πολίτες, ε, αυτό, έχει, αυτό αποτελεί η πολιτική επιλογή, αλλά πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει κάποιο επίπεδο πολυπλοκότητας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Όλαφ ε, λόγω της ε, πολυπλοκότητας ε, επιμένει στην υιοθέτηση εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της απάτης στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη δηλαδή δημιουργούν το απαραίτητο πλαίσιο και περιβάλλον ώστε όλοι οι σχετικοί φορείς να συνεργάζονται για να προστατεύσουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταπολεμήσουν τις ε, απάτης. Εφτά κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει τέτοιες στρατηγικές, ε, άλλα πέντε ε, υιοθετούν αυτή τη στιγμή και άλλα δύο έχουν δεσμευτεί να εκπονήσουν τέτοια στρατηγική. Αυτά λοιπόν είναι ε, θετικά στοιχεία και θα τα δούμε στις εκθέσεις των επόμενων ετών. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια ε, στην εισηγήτρια για την δουλειά της και ευχαριστούμε και τους ευρωβουλευτές για τις παρεμβάσεις τους, τις οποίες θα λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε για την πολύ αναλυτική αυτή και εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Κυρία Τζουφρίντα, θέλετε το λόγο μήπως για να απαντήσετε στις παρατηρήσεις. Να προσθέσω κάποια επιπλέον στοιχεία και ίσως να απαντήσω στις ερωτήσεις που μου έγιναν σχετικά με την ταξινόμηση των κρατών που διαπράττουν τις περισσότερες απάτες ή παρατυπίες Φαίνεται από την έκθεση της Επιτροπής ότι η ταξινόμηση αυτή δεν μπορεί να γίνει γιατί όλα εξαρτώνται από το πότε και πώς ανακοινώνουν τα κράτη-μέλη τις ε, απάτες αυτές. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Υπάρχουν χώρες που μεταφέρουν πολλά τέτοια επεισόδια ενώ άλλες χώρες δεν το κάνουν. Υπάρχουν χώρες που έχουν ε, την διπλή αναφορά και στην Ιταλία συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια ειδική αρχή που δημιουργήθηκε επί τούτου και υπάρχουν και χώρες που δεν το κάνουν καθόλου. Αυτή είναι λοιπόν η δυσκολία της έκθεσής μας. Υπάρχει μια θα έλεγα έλλειψη ενιαίων μεθόδων να αναφέρω την Ιταλία και τη Βουλγαρία μαζί με την Εσθονία είναι πολύ δραστήριες στον τομέα της ανακοίνωσης, της δημοσιοποίησης των απατών. Η Ιταλία τα αναφέρει πολύ συχνά. Ταυτόχρονα κάνει και μελέτες οι οποίες μερικές φορές οδηγούν στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πρόκειται για απάτες αλλά για κάποιες παρατυπίες οι οποίες οφείλονται στην πολυπλοκότητα των διαδικασιών για την απόκτηση των ποσών. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να απαιτήσουμε την περαιτέρω ομογενοποίηση αυτού του συστήματος έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε λίγο τον ορίζοντα και εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία υφίσταται επιθέσεις. Μάλιστα, ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση για το σχέδιο της γνωμοδότησης της κυρίας Τζουφρίντα. Να σας υπενθυμίσω μόνο την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, η οποία τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου στις 12 ώρα το μεσημέρι. Περιμένουμε λοιπόν τις τροπολογίες των συναδέλφων. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Με το επόμενο σημείο στην ομιλητική διάταξη, ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Αναλίζα Μπόνι, Γενική Γραμματέα του Eurocities. Χθες η συνάδελφος Βέστφαλ και Όμπριχτ, Όλμπριχτ μας μίλησαν για την τρίτη συνέλευση του Χάπταρτ στο Κίτο. Θα συνεχίσουμε σήμερα τη συζήτηση για τις μελλοντικές προκλήσεις των ευρωπαϊκών πόλεων με την κυρία Μπόνι, η οποία θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση πρόσφατου έργου του EuroCities θα μας πει ποια είναι η άποψή της για τα αποτελέσματα της τρίτης ε, του τρίτου συνεδρίου του ΧΑΠΤΑ, Θα μας μιλήσει για το αστικό θεματολόγιο και ενδεχομένω θα μπει στον πειρασμό φαντάζομαι να μας αναφέρει τις απόψεις της και για την μελλοντική πολιτική συνοχή, δηλαδή μετά το 2020. Παρακαλώ κυρία Μπόνη, το λόγο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Πρόεδρε, να έχουμε δηλαδή ως γύρω μία ακόμη ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σας. Πράγματι, θεωρούμε ότι τα βασικά θέματα για τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας είναι, η, όπως είπατε, το αστικό θεματολόγιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχατε μια ανταλλαγή για το ΧΑΠΤΑ. Χθε θα κάνω μια διάσυνδεση με το Κίτο και επίσης πράγματι θα υποκύψω και στον πειρασμό όπως είπατε να πω και δύο λόγια για το έργο το οποίο εμείς αυτή τη στιγμή διεξάγουμε για την πολιτική συνοχή με το 2020. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το αστικό θεματολόγιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε όλοι, ήσασταν και κάποιοι από εσάς εκεί, γνωρίζουμε όλοι ότι το σύμφωνο του Άμστερνταμ εγκρίθηκε την 30η Μαΐου στο Άμστερνταμ βέβαια, 20 χρόνια δηλαδή μετά από συνομιλίες και συζητήσεις. Έχουμε λοιπόν πλέον ένα αστικό θεματολόγιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά δεν πρόκειται για ένα ενωσιακό θεματολόγιο ή μια ενωσιακή πολιτική. Όμω είναι ένα πολύ καλό σημείο αφετηρία, κατά την άποψή μου, ώστε να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εργάζεται καλύτερα για και με τι πόλει, για τι συγκεκριμένε προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τι οποίε εσεί αποφασίζετε και εμεί βέβαια επί τόπου. Οι βασικέ προκλήσει λοιπόν που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το θέμα. Θέλω να σα υπενθυμίσω ότι οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα επικεντρώνουν ουσιαστικά, εστιάζονται τι πόλει. Κλιματική αλλαγή, φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό, ανεργία, προσφυγική κρίση. Πρόκειται στο σύνολό του για προκλήσει και ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλει σε καθημερινή βάση. Όπως γνωρίζετε λοιπόν το θεματολόγιο εστιάζει σε 12 θέματα και προτείνει ορισμένα εργαλεία όπως είναι οι εταιρικέ σχέσεις, θεματικές εταιρικέ σχέσεις. Είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω του αστικού θεματολογίου. Βέβαια, πρόκειται για τις απαρχές, εφόσον εγκρίθηκε μόλις το Μάιο αυτό το θεματολόγιο, συν κάποιε από τις εταιρικέ σχέσεις που ξεκίνησαν πριν από 9-10 μήνες. Όμως, θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να έχουμε εδώ μια συζήτηση για ορισμένα ζητήματα. Ποια είναι τα καλά πρώτα. Παραλαμβάνω, το αστικό θεματολόγιο, η ύπαρξή του και μόνο, είναι ένα τεράστιο αποτέλεσμα αυτό το σύμφωνο, ένα τεράστιο ε, θετικό αποτέλεσμα. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ έχει βοηθήσει, έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, όπως πάντοτε. Επίσης η Ολλανδική Προεδρία έδωσε μεγάλη όθηση και εσείς στήριξατε με τις εκθέσεις πρωτοβουλίας και άλλους τρόπους αυτό το θεματολόγιο όπως και εμείς έχουμε λοιπόν πλέον αυτό το θεματολόγιο συλλογική προσπάθεια σε θεσμικό επίπεδο και επίπεδο αστικών ε, κέντρων ήταν πάρα πολύ μεγάλη αυτή η προσπάθεια και έτσι πρέπει να παραμείνει και του επόμενου μήνες και χρόνια δυνατόν τέσσερα πιλωτικά Τέσσερι πιλωτικέ εταιρικέ σχέσει έχουν ήδη ξεκινήσει για την ποιότητα του αέρα, τη στέγαση, τη μετανάστευση και τι ήτανε. Α, τη φτώχεια. Αυτά είναι τα τέσσερα. Αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει. Και ήδη βλέπουμε κάποια αποτέλεσμα. Δεν ήταν εύκολο. Αυτό μπορώ να σας το πω. Γιατί να κάτσουν στο τραπέζι πόλης, ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και κομισιόν για αυτά τα θέματα, να συζητήσουν και να βρουν κοινό έδαφος και να αποφασίσουν ότι ναι αυτό ή το τάδε ή το δίνα θέμα θα το αντιμετωπίσουμε, ξέρετε ότι όλα αυτά απέτησαν μεγάλη προσπάθεια από όλους. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένε ιδέες οι οποίες ξεκινούν πλέον να αποκρισταλώνονται. Θα αρχίσει να πιάνει η μαγιονέζα σιγά σιγά. Sorry. Now, there is a... Επίσης οι πόλεις έδειξαν πάρα πολύ θετική ανταπόκριση και αυτό δεν ήταν δεδομένο στην αρχή. Λέγαμε αρχικά πώς μπορούν και οι πόλεις να ενδιαφερθούν, να επενδύσουν πόρους, ε, να συμμετάσχουν σε αυτές τις εταιρικές σχέσεις και το καθεξής. Όμως τελικά βλέπουμε ότι οι πόλεις ε, ανταποκρίνονται σε πάρα πολύ ε, μεγάλο βαθμό. Να μην πω ότι έχουν πάθει ψύχωση και θέλουν να καθίσουν σώνη και καλά στο τραπέζι αυτών των διαπραγματεύσεων γιατί η τάδε πόλη και όχι η δική μου και ούτω Τέτοια πράγματα βλέπουμε. Το τρίο των προεδριών, οι τρεις προεδρίες ε, και η Κομισιόν ε, κατάφεραν ε, να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πόλεων, άρα των κρατών μελών δηλαδή, αλλά και έχουν δώσει την έμφαση εκεί που τα μηνύματα θα μπορούσαν να δοθούν από περισσότερες πόλεις ως δίκτυα. Εκτός του πίνακα, αν θέλετε, των εταιρικών σχέσεων. Οι πέντε πόλεις που θα καθίσουν ε, στο τραπέζι γύρω από την ίδια σχέση θα είναι κατά κάποιο τρόπο εκπρόσωποι μιας μεγαλύτερης κοινότητας και θα μπορούν να μεταφέρουν σημαντικά μηνύματα που μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγέ. Ένα άλλο θετικό σημείο είναι ότι ήδη έχουμε του συντονιστέ για τι επόμενε τέσσερι εταιρικέ σχέσει και οι πόλει που έχουν επιλεγεί ήδη για τι επόμενε εταιρικέ σχέσει και στα μέσα του επόμενου έτου θα έχουμε τι άλλε τέσσερι. Άρα, μέχρι τα τέλη του 2017, αν δεν κάνω λάθο, θα έχουμε του 12 πίνακε και θα έχουμε έτοιμε τι 12 εταιρικέ σχέσει σε ό,τι αφορά την τεχνική βοήθεια και την υποστήριξη. Ε, προκήρυχθηκαν οι σχετικοί διαγωνισμοί, υπάρχουν και τα, υπήρξε και το πιλωτικό πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά θα έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, καλά όλα αυτά, όμως, νομίζω ότι είναι σημαντικό η προσοχή να παραμείνει και σε κάποιες άλλες πτυχές. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να διατηρήσουμε ε, το ρυθμό και να βελτιώσουμε ήδη ε, και αν ή δυνατόν αυτό το έργο που έχει ξεκινήσει. Θέλουμε αυτό το σύμφωνο να κάνει τη διαφορά για τις αστικές πολιτικές. Άρα θα πρέπει να δούμε ορισμένα θέματα. Κατά την άποψή μας τα σημαντικά θέματα είναι πρώτο. δεν υπάρχει ακόμη επαρκή δέσμευση εκ μέρους των κρατών μελών. Είναι ένα σύμφωνο όμω αυτό μεταξύ των κρατών μελών. Όχι με τι τα κράτη-μέλη. Οι υπουργοί αστική ανάπτυξη τα συμφώνησα. Δεν βλέπουμε όμω και πολλού να κάθουν στο τραπέζι των εταιρικών σχέσεων. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να υπάρξει ε, έργο και σε εθνικό επίπεδο. Εμεί ε, στο πλαίσιο του EuroCities και φαντάζομαι και στο επίπεδο κοινοβουλίων γίνεται προσπάθεια να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από τα κράτη-μέλη. Αλλιώ δεν έχει και νόημα να υπάρχουν εταιρικέ σχέσει στι χώρε μέλη που δεν ενδιαφέρονται Τώρα με τις τομιακές γαμαδέλτα της Κομισιόν τα πράγματα βελτιώνονται. Ίσως όμως χρειαστεί πέραν της γαμαδέλτα Ρέτζιο που αυτή πιέζει πιο πολύ και βάζει τη, κάνει το μεγαλύτερο προσπάθεια και άλλες τομιακές γενικές διευθύνσεις. Παραδείγματο χάρη συζητάμε οδηγίες για την ποιότητα του αέρα. Δεν χρειάζεται και το περιβάλλον καθίσει στο τραπέζι. Πάντοτε με την υποστήριξη από το συντονισμό της γαμαδέλτα βέβαια όπως είπα, κάνει τη μεγάλη προσπάθεια και δίνει την όθηση. Αλλά χρειάζονται και οι άλλες σχετικές γενικές διευθύνσεις. Γάμα δελτα ανταγωνισμός, παραδείγματος χάρη συνεταιρική σχέση για τη στέγαση. Κρατικές ενισχύσεις για τις προσιτές κατοικίες. Το είδαμε ότι πρέπει να κάθονται οι άνθρωποι αρμόδιοι και οι υπουργοί και οι τομεακές γενικές διευθύνσεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί και στο επισημαίνουμε. Σας το επισημαίνουμε. Δεύτερο στοιχείο που επισημαίνουμε. Πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή για να παραμείνει το ενδιαφέρον σε αυτό το θέμα. Φυσικά και δεν είναι ε, δεσμευτικό, δεν αναφέρεται στη συνθήκη το σύμφωνο, είναι το περισσότερο μπορέσαμε να πετύχουμε. Πώς όμως θα εγγυηθούμε, πώς θα εξασφαλίσουν και εγώ ε, με τη διαδικτύωση μέσω του EuroCities, πώς θα κρατήσω ε, το Δήμο μου, την πόλη μου ε, να ενδιαφέρεται. Πώς θα διατηρήσω το ενδιαφέρον, αν δεν τροφοδοτούνται τις ευρωπαϊκές διαδικασίες, την νομοθετική και άλλες, τα αποτελέσματα των εταιρικών σχέσεων. Θα μπορέσουν οι εταιρικές σχέσει αυτές να αλλάξουν τα πράγματα όταν αυτά δεν λειτουργούν. Να λύσουν κάποιες συμφορήσεις ό,τι αφορά παραδείγματο χάρη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Επιτόπου και πώς εφαρμόζεται. Αυτό για μας είναι σημαντικό. Στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2017 ούτε μια λέξη δεν υπάρχει για τις πόλεις. Ούτε καν η λέξη πόλη δεν αναφέρεται. Αλλά όλα αυτά τα οποία αναφέρει το πρόγραμμα εργασίας της πόλης λαμβάνουν χώρα. Είναι ένα στοιχείο που μας ανησυχεί λοιπόν. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχει μια καλύτερη διασύνδεση με τις νομοθετικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, καλύτερη νομοθεσία. Πώς θα συσχετίσουμε το θεματολόγιο αυτό. Ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς πώς θα συμμετάσχει περισσότερο και επίσημα σε αυτή τη διαδικασία για να διαπιστωθεί ότι πράγματι μπορούν να προκύψουν από αυτές τις εταιρικέ σχέσεις ιδέες για τη βελτίωση τη νομοθεσία και να ληφθούν υπόψη. Το θέμα δηλαδή είναι ουσιαστικά να διατηρηθεί η πολιτική, θεσμική όθηση και ορμή για τους επόμενους μήνες και χρόνια. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο, σημαντικό μάλιστα ρόλο, να παρακολουθεί να ελέγχει και να βλέπει ότι όλες οι προσπάθειες, όλο το έργο αυτό που γίνεται συλλογικά, ομαδικά και από θεσμικής πλευράς αλλά με τις κοινότητες, αλλά και τα πορίσματα, οι μεθοδολογίες, τα αποτελέσματα των εταιρικών σχέσεων, θα πρέπει, όπως είπα, να τροφοδοτούν τη διαδικασία λήψος αποφάσεων. Πολύ συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι και η Επιτροπή Ρέγγι και τα μέλη της Επιτροπής σας έχουν ρόλο, αλλά και το, η αστική ομάδα εργασία, το Intergroup για τα αστικά θέματα. Θα πρέπει να παρακολουθείτε και από πολιτικής πλευράς σε καθημερινή βάση το έργο των εταιρικών σχέσεων. Το Urban Intergroup θα μπορούσε να προσκαλέσει τις πόλεις για παράδειγμα. Τους συντονιστές, της κομισιόν και συγκεκριμένες πόλεις που συμμετέχουν στη διαχείριση των εταιρικών σχέσεων για να σας ενημερώσουν για το έργο τους. Και να δείτε κι εσείς τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί, πώς μπορεί να βοηθήσει το input αυτό και τις χώρες μέλη. Ή θα μπορούσε η Επιτροπή σας να αξιοποιήσει τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τι εταιρικές σχέσεις για τον προβληματισμό σας σε σχέση με τη μελλοντική στρατηγική ε, και πολιτική συνοχή μετά το 2020. Και εδώ μπαίνω στον περιορισμό να σας κάνω κάποιες προτάσεις για την πολιτική συνοχή σε σχέση με τις συνέργειες ε, που υπάρχουν για μετά το 2020. Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω το εξής. Πώς μπορούμε τα αποτελέσματα των εταιρικών σχέσεων να τα αξιοποιήσουμε, να τα αξιοποιήσετε εσείς στον προβληματισμό σας και στη γενική σας συλλογιστική πάνω στη μελλοντική πολιτική συνοχή Για τα θέματα πρώτα απ' όλα. Πρόσφυγες, μετανάστευση, όλα αυτά τα θέματα έχουν να τα αντιμετωπίσουν σίγουρα πολύ έντονο τρόπο οι δήμαρχοι, οι πόλει. Και στην τρέχουσα περίοδο έγιναν απόπειρε αλλαγή του επιχειρησιακού προγράμματο. Δεν είναι εύκολο αυτό όμω. Ένα παράδειγμα που μπορώ να δώσω είναι οι βασικέ προκλήσει που αντιμετωπίζονται μέσω των εταιρικών σχέσεων. Πώ θα μπορούσαν να επηρεάσουν τι πολιτικέ προτεραιότητε τη πολιτική συνοχή. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, πώ μπορούμε να μπούμε στις λεπτομέρειες, να δείξουμε με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει ότι υπάρχουν ανάγκες των πόλεων οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν ε, την, τη μεγαλύτερη κατανόηση και πώς οι πόλεις συμμετέχουν στο σχεδιασμό των προτεραιοτήτων. Πόσο συμμετέχουν οι πόλεις ε, στην, ε, στον εντοπισμό των τοπικών αναγκών, στον καθορισμό των τοπικών αναγκών που θα πρέπει να καλύψει και να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα. Και έρχομαι στο δεύτερο σημείο για την πολιτική συνοχή που είναι η αρχή της εταιρικής σχέσης. Το αστικό θεματολόγιο δείχνει και βασική αρχή, βασική λογική έχει αυτήν την προσέγγιση της εταιρικής σχέσης. Κράτη-μέλη, κομισιόν, πόλης, κοινοβούλιο, όλοι αυτοί οι θεσμοί συνεργάζονται για να δώσουν αποτέλεσματα επιτόπου ό,τι αφορά τι βασικέ ενωσιακέ προτεραιότητε. Αυτό πρέπει να γίνει. Και θα πρέπει και η πολιτική συνοχή να ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο. Μέχρι στιγμής δεν ήταν ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. Αν δείτε τον κώδικα συμπεριφορά σε ό,τι αφορά την αρχή σχέση, πάνω στο χαρτί μια χαρά είναι όλα γραμμένα. Τι κάνουν όμω στην πράξη. Δεν συμμετέχουν στι διαβουλεύσει οι πόλει για την επιλογή προτεραιοτήτων, για τη διαχείριση, την υποστήριξη, για τη χρήση των κονδύλιων συνοχής στι περιοχέ του. Πολλά μπορούμε να κάνουμε από κοινού και χρειαζόμαστε και τη δική σας υποστήριξη για να εφαρμόσουμε την αρχή της εταιρική σχέσης και στα διαθετικά ταμεία για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού με πολύ μεγαλύτερη έμφαση. Διότι βλέπουμε όλοι ότι η κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη σχετίζεται με το ότι απέχει πολύ η Ευρώπη από το τοπικό επίπεδο, τους πολίτες. Όλοι συμφωνούν από αυτού. Πώς μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε την πολιτική συνοχή για να έχουμε ένα πιο μεγάλο σύνδεσμο και δεσμό με... Οι προτεραιότητες τώρα. Η αρχή της εταιρικότητας και τα ολοκληρωμένα μέσα τα οποία πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας, τα εδαφικά μέσα. To deliver the funds in an integrated way, these are also important tools that Όλα αυτά δεν ε, μπόρεσαν ε, να τα εφαρμόσουν αρκετά στο πρόγραμμα αυτής της περίοδου. Το θέμα είναι πώς μπορούμε λοιπόν να τα βελτιώσουμε αυτά και να έχουμε τα απλοποιημένα ITI ε, ικανά να συνεργαστούν μεταξύ τους και να καταλήξουμε σε καλύτερες λύσεις. Νομίζω ότι είναι προς όφελος όλων να υπάρχει μια καλύτερη σε εισαγωγικά παράδοση των ε, διαφθρωτικών ταμείων ε, ε, επιτόπου. Είδατε τα αποτελέσματα των καινοτόμων ενεργειών στον τομέα των αστικών περιοχών. Οι πόλεις ανταποκρίθηκαν με ικανοποίηση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε και εμείς με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε τα διαφθρωτικά ταμεία και τις καινοτόμες ενέργειες. Οι πόλεις ε, είναι ε, ικανές να το κάνουν. Έχει σημασία οι εθνικές διαχειριστικές αρχές και οι περιφερειακές αρχές να αναγνωρίσουν ότι οι πόλεις μπορούν να δεχθούν τις παρεμβάσεις αυτές. Ίσως όχι όλες με τον ίδιο τρόπο, κάποιες να χρήζουν περισσότερης ε, τεχνικής βοήθειας όχι μόνο σε επίπεδο διαχείρισης του Ταμείου αλλά και της ε, επιτόπου ανάπτυξης ε, του Ταμείου. Αλλά πάντως νομίζω ότι μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχουν μερικές φορές κάποια, κάποια εμπόδια από πλευράς εθνικών αρχών διαχειριστικών και τοπικών διαχειριστικών αρχών. Δεν είναι οικονομικό το θέμα, δεν μπορούμε να τους δώσουμε περισσότερα χρήματα γιατί δεν θα τα καταφέρουν. Και τέλος υπάρχει και το θέμα της απλοποίησης, πάνω σε αυτό ακούστηκαν αρκετά προηγουμένως. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε. Είμαι μέλος της ομάδας υψηλού επίπεδου για την απλούστευση των διαδικασιών Νομίζω ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν στο να γίνει η πολιτική μας πιο αποτελεσματική, πιο απλή και σε σχέση με τις κρατικές επιδοτήσεις και σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες. Πρέπει να συγχρονίσουμε τις προσπάθειες, εδώ υπάρχει και ο δικός σας ρόλος. Οι κανονισμοί διαθέσιμοι θα πρέπει να αναλυθούν και να εγκριθούν πολύ νωρίτερα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο η έκθεση ε, ε, για την συνοχή θα ε, δοθεί στο τέλος του 2017. Αυτό αποτελεί ένα κίνδυνο διότι δεν θα επιτρέψει την σωστή εκτέλεση των προγραμμάτων. Λοιπόν, αυτά για την πολιτική συνοχή. Πάντως θα ήθελα να πω ότι το τελικό μας, λέω τώρα, μήνυμα προς εσάς είναι ότι απαιτείται να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρώπη τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε δεκτικοί και να μπορέσουμε να επαναπροσανατολίσουμε την συζήτηση. Αυτό ζητούν οι τοπικοί μας άρχοντες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε την απόσταση ανάμεσα στα επίπεδα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τον πολίτη. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι σημαντικό και θα πρέπει να εφαρμοστεί από όλους. Το θέμα είναι όμως να εμπλέξουμε τις τοπικές αρχές, να τους ακούσουμε, να συνεργαστούμε μαζί τους. Αυτή είναι η προτεραιότητα του δικού μας δικτύου και ακριβώς η ατζέντα για τις αστικές περιοχές είναι, έχει αυτό το πνεύμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει ε, να μην υπάρξει άλλο Brexit. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε εθνικιστικά κινήματα και αντιευρωπαϊκά κινήματα να συνεχίσουν να αναπτύσσονται θέλουμε να είμαστε σύμμαχοί σας στην διαδικασία αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι θα πρέπει να απευθύνουμε μια έκκληση για να υπάρξει μια συμμαχία για την αναθεώρηση της Ευρώπης, για την επανασύνδεση της Ευρώπης με τις πόλεις μας. Την 7η Μαρτίου του 2017 θα έχουμε μια συνάντηση κορυφής δημάρχων έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή και με τις ηγεσίε των χωρών να δούμε πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε έναν δρόμο θετικό και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι λιγάκι λιγότερο καταθλιπτικό από το παρόν και να έχουμε έτσι μια πιο ισχυρή Ευρώπη αντίθετα από την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε σε αυτή την συνάντηση κορυφής, να συνεργαστούμε ε, μαζί σας. Τώρα για το Κίτο δεν θα μιλήσω, είχατε τη συζήτηση χθε. Είπα ότι δεν θα μιλήσω, αλλά παρόλα αυτά η σύνδεση ανάμεσα στην ατζέντα του Κίτο και την δική σας ε, είναι κάτι το οποίο και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε υπηρετικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σαφές ότι τα προβλήματα τα βασικά είναι στις πόλεις. Υπάρχει ανάγκη οι πόλεις να είναι υποσυζήτηση. Οι προκλήσεις των πόλεων είναι ακριβώς το θέμα και εκεί θα βρούμε και τις λύσεις. Νομίζω λοιπόν ότι μια τέτοια προσπάθεια θα ενισχύσει και τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της ατζέντα αυτής για τις αστικές συγκεντρώσεις και οι συνέργειες σε διεθνές επίπεδο θα βοηθήσουν. Τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν ε, την ε, ομιλία θα παρακολουθήσουμε τις εργασίες σας, διότι θα είναι ενδιαφέρον ε, για τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζη να δουν τι συμβαίνει. Θα ανοίξω τη συζήτηση. Κυρία Μπρέσο, θέλετε τον λόγο, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αναλίζα Μπόνη και τις υπηρεσίες της για αυτήν την εμπνευσμένη ανάλυση την οποία μας έκανε για την κατάσταση, για τα θέματα των πόλεων για τον ρόλο των πόλεων στην πολιτική συνοχής και στις ευρωπαϊκές πολιτικές γενικότερα. Εμείς με αυτά ασχολούμεθα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το θέσουμε για συζήτηση. Θα συμφωνήσω λοιπόν και δεν θα μακρηγορήσω για την ανάλυση την οποία κάνατε. Πράγματι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πόλεις ε, είναι αυτές οι οποίες ε, λαμβάνουν τα περισσότερα κοινοτικά διαφορετικά κονδύλια. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν η ζήτηση, το αίτημα είναι να εμπλακούν ακόμα περισσότερο ε, στο επίπεδο του συνολικού προγραμματισμού της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μπορέσουν να ορίσουν καλύτερα τους όρους οικοδόμησης της στρατηγικής αυτής και να συμμετέχουν στην, στην ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών και να προσφέρουν την δική τους εμπειρία λοιπόν και την δική τους ικανότητα δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών στις αστικές συγκεντρώσεις. Εγώ και ως πρόεδρος ενός intergroup για το υπόλοιπο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τις περιφερικές και ορεινές περιοχές, έχω φυσικά ασχοληθεί και με τις αστικές περιοχές, εγώ η ίδια μένω σε πόλη και επίσης θα έλεγα ότι αγαπώ και τις πόλεις, αλλά εν πάση περιπτώσει Νομίζω ότι οι εκπρόσωποι των οργανώσεων των πόλεων επιτρέπουν στα πλαίσια των προτάσεων τους στο εσωτερικό της πολιτικής συνοχής και στα πλαίσια της συγκέντρωσης των στόχων και του mainstreaming της Ευρώπης 2020 με τις άλλες προτεραιότητες αυτή η καλή προσπάθεια δεν θα πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε ότι τα κοινοτικά εδάφη είναι πολυπίκυλα, ότι οι ορινές περιοχές έχουν κάποιες προτεραιότητες διαφορετικές από τις αστικές περιοχές. Διερωτώμε λοιπόν αν την επόμενη προγραμματική περίοδο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το εξής. Για το θέμα της συγκέντρωσης των παρεμβάσεων να ξεκαθαριστούν οι προτεραιότητες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των περιοχών και εδαφών. Δηλαδή, δεν είναι αλήθεια ότι ένα πρόγραμμα καλό ισχύει για όλους Νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι καλό για όλους είναι ο σωστός προγραμματισμός και ο σωστός καθορισμός των προτεραιοτήτων. Αν ας πούμε προτεραιότητα είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Αυτό είναι σαφές. Από την άλλη, οι ανάγκες είναι διαφορετικές στα βουνά ή στις πόλεις. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε την διαφοροποίηση που απαιτείται. Κατά τα άλλα, η εμπειρία των γεροσύτης θα είναι πολύτιμη για τις εργασίες μας, για την επόμενη νομοθετική ρύθμιση και για τις επόμενες στρατηγικές που θα ακολουθήσουμε. Γιατί θεωρώ ότι πολλά από τα κατεπήγοντα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σωστά παρά μόνο μέσω μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης με τις πόλεις. Υπάρχουν προβλήματα βέβαια κυρίαρχα όπως το μεταναστευτικό που σίγουρα θα αντιμετωπιστούν κυρίως μέσω των πόλεων. Ευχαριστώ λοιπόν. Περιμένουμε και γραπτές προτάσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξανασκεφτούμε τις προτάσεις σας και κάτι το οποίο συζητήσαμε και προηγουμένως είναι ότι όπως είπατε ανήκετε στην ομάδα απλοποίησης θα θέλαμε από πλευρά σας συγκεκριμένες παρατηρήσεις, προτάσεις για τις απλουστεύσεις όχι μόνο μέσα από τις εμπειρίες τις οποίες συλλέγετε στην ομάδα που συμμετέχετε αλλά να μα τις στείλετε σε εμά τις εμπειρίες και τις προτάσεις σας είναι χρήσιμο να τις έχουμε υπόψη τις προτάσεις των πόλεων γιατί οι πόλεις είναι οι βασικοί διαχειριστές των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ε, ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Μπόν για την παρέμβασή της. Θέλω και εγώ ένα παρόμοιο ερώτημα να θέσω με αυτό τη συναδέλφου, δηλαδή συγκεκριμένα. Η EuroCities ε, ποια θέση έχει για την απλούστευση. Είναι ένα θέμα επίκαιρο, το συζητούμε στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα λοιπόν το EuroCities να μας πει και η ομάδα υψηλού επίπεδου σε ποιο επίπεδο βρίσκεται σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και τις συστάσεις. Ε που θα διατυπώσει. Και τι ζητά το EuroCities ε, στο πλαίσιο αυτού του έργου. Thank you. Other wishes for... Ευχαριστώ. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να κάνει παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι αρμόδιο για το αστικό θεματολόγιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι πολύ με τα όσα άκουσα από την Ανάλυζα Μπόνη. Ε, συμμεριζόμαστε τις περισσότερες από τις θέσεις της. Ε, λίγες παρατηρήσεις σε απάντηση των όσων είπε. Καταρχάς, όσον αφορά το ρόλο των κρατών μελών, είναι αλήθεια ότι ε, στις ε, πρώτες ε, τέτοιες σχέσεις δεν είχαμε αρκετά τα κράτη-μέλη για τις τέσσερις πρώτες. Ε, για τις επόμενες όμως είχαμε υπερβολικά πολλά και έπρεπε να περιορίσουμε την ε, συμμετοχή τους. Ε, θα έχουμε λοιπόν αρκετά κράτη-μέλη στο μέλλον. Τα κράτη-μέλη επίσης συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ομάδας για την αστική ανάπτυξη και καλούμε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τις συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων Υπουργείων και των διαφόρων χωρών. Τα κράτη-μέλη λοιπόν ε, έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη έχει να κάνει με την ε, συμμετοχή, με την ε, ναι, με την ε, συμμετοχή των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, είναι σαφές ότι ε, αυτές που έχουν να κάνουν με τα θέματα αυτά θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά ακόμα και αν δεν είναι επικεφαλής. Για παράδειγμα, όσον αφορά την κυκλική οικονομία θα πρέπει να συμμετέχει η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος αλλά και ανάπτυξης, ανταγωνισμού και πολλές άλλες γενικέ διευθύνσει. Ε, για παράδειγμα, εταιρική σχέση για την ποιότητα του αέρα. Έχουμε δύο γενικέ διευθύνσει ε, την ε, περιβάλλοντο και ενέργεια που είναι μέλη. Έχουμε όμω και μια ομάδα όπου συμμετέχει η Γενική Διευθυνσή μου, η Grow, η έρευνα, που συμμετέχουν στις προπαρασκευαστικές εργασίες. Καταβάλουμε λοιπόν κάθε προσπάθεια. Ε, αποτελεί στόχο μας και συμφωνούμε απολύτως ότι χωρίς ε, την ε, συμμετοχή τους η ποιότητα των εταιρικών σχέσεων δεν θα είναι όσο καλύτερη γίνεται. Τρίτη παρατήρηση, η εγγύηση ότι οι εργασίες ε, του αστικού θεματολογίου και των ε, εταιρικών σχέσεων θα είναι χρήσιμοι. Φυσικά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, διότι είναι ακόμα πολύ νωρίς, ε, αλλά μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι θα εξετάσουμε τις συστάσεις. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα εφαρμοστούν όλες οι συστάσεις, υπάρχει όμως η εγγύηση ότι θα εξετάσουμε το σχέδιο δράσης και όταν λέμε εμείς, ενώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά κυρίως οι συνομοθέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Έχετε λοιπόν και εσείς σημαντικό ρόλο να παίξετε. Γι' αυτό τέθηκε και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με φέρνει στην τέταρτη μου παρατήρηση. Είναι σημαντικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο σύμφωνο του Άμστερνταμ αναφέρεται ρητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει να παίξει πραγματικό ρόλο. Επίσης είναι προσκεκλημένη ε, οι αρμόδιοι άνθρωποι και πάντα ανταποκρινόμαστε στις προσκλήσεις από δική σας πλευράς. Ε, αν οι συστάσεις έχουν να κάνουν με την τροποποίηση μιας οδηγίας ε, ή κάποιου δημοσιονομικού μέσου, τότε κυρίως ε, αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του νομοθέτη και όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο λοιπόν είναι σημαντικοί παράγοντες για να είναι χρήσιμη, χρήσιμο το αστικό θεματολόγιο. Τελευταία μου παρατήρηση για την πολιτική συνοχής. Καταλαβαίνουμε τις δυνατότητες του αστικού θυματολογίου και τις συστάσεις για το επόμενο διάστημα για την επόμενη περίοδο της πολιτικής συνοχής ε, και γι' αυτό ε, συστήσαμε όσους εργάζονται πάνω στο θέμα αυτό να εξετάσουν πρώτα αυτό ώστε οι σχετικές συστάσεις να φτάσουν εγκαίρως να μην χρειάζεται δηλαδή να συλλέξουμε όλες τις συστάσει για το σχέδιο δράσης προτού να ξεκινήσουμε τις εργασίες, ε, να μπορούμε να ξεκινήσουμε την εργασία σε φάσεις, δηλαδή πρώτα τα πιο επίγοντα ε, και σε δεύτερη φάση άλλα θέματα. Αυτά λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον προπολογισμό που μα διαθέσατε, που θα χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία γραμματεία. και αυτό θα βοηθήσει πολύ την ε, διαχείριση του αστικού θεματολογίου. Σας ευχαριστούμε και πάλι λοιπόν. Και το, ξανατονίζω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και πάντα είμαστε στη διάθεσή σας για να σας δώσουμε στοιχεία κλπ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Μπόνη, έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις ε, που ακούσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. μία παρατήρηση για αυτό που είπε η Μεσέντες σχετικά με τις ε, συνέργειες ε, ε, αστικού και υπαίθριου επίπεδου. Πολύ ευχαριστώ θα εξετάσουμε αυτές τις συνέργειες και θα τις συζητήσουμε περαιτέρω. Σκεφτόμαστε να εξετάσουμε και την μητροπολιτική διάσταση των μεγάλων πόλεων, διότι πολύ συχνά αυτές οι περιοχές των μεγάλων πόλεων περιλαμβάνουν και ε, πιο υπαίθριες ε, περιοχές ε, και τίθεται το θέμα της κινητικότητας ανάμεσα στις περιοχές αυτές. Όπως επίσης η αγορά εργασίας είναι θέμα που μας ενδιαφέρει εδώ. Θέλουμε λοιπόν μια περισσότερο εις βάθος συζήτηση για τα θέματα αυτά και πολύ ευχαρίστως θα σας στείλουμε γραπτές παρατηρήσεις. όσον αφορά το αίτημα για την ε, ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλούστευση και την ε, κατάσταση όσον αφορά την ομάδα αυτή. Τέσσερις εκθέσεις έχουν εκπονηθεί, μία για τα δημοσιονομικά μέσα, για να βελτιωθεί η χρήση των εργαλείων αυτών, μία για ε, τις απλουστευμένες δαπάνες, διότι αυτό αποτελεί μέρος του ισχύοντος κανονισμού. Δεν εκμεταλλευόμαστε όμως αρκετά αυτή τη δυνατότητα, επειδή υπάρχουν φόβοι, έλλειψη εμπιστοσύνη στον δικαιούχο, ή στις αρχές διαχείρισης όσον αφορά τη δυνατότητά τους ε, να ε, συμμορφώνονται με τους κανόνες ε, όσον αφορά το λογιστικό έλεγχο κλπ. Υπάρχουν λοιπόν πολύ συγκεκριμένες συστάσεις. Πολύ συγκεκριμένες συστάσεις επίσης στην έκθεση για το θέμα της πρόσβασης από πλευράς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πώς μπορούμε να την βελτιώσουμε. Και τελευταία τελευταίο θέμα στο οποίο ήμουν συνεισηγήτρια μαζί με ε, πολλοί ευρωβουλευτή είναι ο, ο ε, κανονιστικός υπερθεματισμός, το gold plating. Αυτή μάλλον είναι και η πιο ευρεία έκθεση, διότι εξετάζει όλα τα θέματα που αποτελούν ε, πηγή ε, προβλημάτων για τις περιφερειακές αρχές, ε, τις εθνικές αρχές κλπ. Και εξετάζει τι σημεία συμφόρησης υπάρχουν, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα διαστοτικά ταμεία, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα μέτρα απλούστευσης που προβλέπονται και όλα αυτά. Στόχο είναι λοιπόν στην έκθεση αυτή να δείξουμε ότι ο κανονιστικό υπερθεματισμός που γενικά θεωρείται η υπερβολική νομοθεσία από πλευράς των εθνικών και υποεθνικών αρχών αυτή η κατάσταση δημιουργείται και λόγω της ε, Ε, πολυπλοκότητας των εθνικών κανόνων και της μεταφοράς τους στο εθνικό δίκαιο. Δεν φταίνε λοιπόν αποκλειστικά οι εθνικές αρχές. Η πολυπλοκότητα, η δυσκολία της συμμόρφωσης με όλα αυτά τα επίπεδα νομοθεσίας βάζουν σε δύσκολη θέση τις διαχειριστικές αρχές. Και ένα από τα στοιχεία που έχει επισημανθεί ε, στην εκθεσή αυτή είναι το θέμα του λογιστικού ελέγχου, διότι πολλές από αυτές τις αρχές διαχείρισης δεν εφαρμόζουν τη δυνατότητα απλοποιημένων δαπανών, διότι φοβούνται ότι κατά το λογιστικό έλεγχο δεν ε, θα μπορούν να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς που είναι πολύ αναλυτικοί. Οι εθνικές ε, και περιφερειακές αρχές λοιπόν ε, θέλουν να προστατευτούν και γι' αυτό νομοθετούν υπερβολικά. Ο λογιστικός έλεγχος λοιπόν ε, θεωρήθηκε σημαντικό πρόβλημα τομέας όπου χρειάζεται απλούστευση και από τον Όλαφ μέχρι το περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει ελέγχονται μάλλον τα ίδια προγράμματα κλπ. Αλλά θα πρέπει να έχουμε προσέγγιση με βάση την αρχή της επικουρικότητας, ώστε το ευρωπαϊκό επίπεδο να ελέγχει τα συστήματα ελέγχου και την ποιότητά τους σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να πρέπει να μπουν σε λεπτομέρειες συγκεκριμένων προγραμμάτων που θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα του εθνικού και υποεθνικού επίπεδο, επίπεδου, ώστε να μην έχουμε υπερβολικά πολλούς λογιστικούς ελέγχους και οι δικαιούχοι ε, να μην αντιμετωπίζουν αυτό το άχθος. Δηλαδή, ακόμα και για ε, κάτι που στοιχίζει 10 ευρώ γίνεται ο, ο λογιστικός έλεγχος σε 5 επίπεδα. Κατόπιν έχουμε το θέμα των κρατικών ενισχύσεων ε, και των ε, κανόνων ε, που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. Πρόκειται για θέματα που ρυθμίζονται πολύ αναλυτικά, ώστε να έχουμε περίπου χίλιες σελίδες που πρέπει να μάθουν να μελετήσουν οι, δημόσιες, οι διαχειριστικές αρχές ε, αλλά και κάθε μικρή επιχείρηση. Θα πρέπει λοιπόν κάθε μικρή επιχείρηση να δει πώς ε, να αντιμετωπίσει τα διάφορα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν είναι αδύνατο να γίνει. Συγκεκριμένη σύσταση λοιπόν, ε, όταν εγκρίνονται τα επιχειρησιακά σχέδια, να εγκρίνεται και το καθεστώς δημοσίων συμβάσεων, ώστε κατά τη διάρκεια της επταετίας να μην πρέπει να προσφεύγει κανείς σε συνέχεια στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Όταν κλείσει το πρόγραμμα λοιπόν να έχει κλείσει και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να είναι ικανοποιημένη με αυτό. Αλλά βέβαια αυτό είναι πολύ πολιτικό θέμα διότι έχει να κάνει με την πολιτική ανταγωνισμού. Οι κρατικές ενισχύσεις ε, είναι μία από τις πιο σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πάντως, εμείς έχουμε υποβάλει πολύ συγκεκριμένε συστάσεις για το θέμα αυτό. Το ίδιο ισχύει για την ε, δευτερογενή νομοθεσία ε, με το παράγωγο δίκαιο. Έχετε, λοιπόν, το δικό σας παράγωγο δίκαιο στο οποίο έχετε συνομοθετήσει, το RDF, τον Γενικό Κανονισμό, για το ESF κλπ. Μάλλον αυτή, αυτό είναι το κύριο δίκαιο, αλλά υπάρχουν κατόπιν ε, πολλά, ε, πολλές πράξεις ε, του παράγωγου δικαίου που δημιουργούν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο ε, νομοθετικό περιβάλλον για όσους πρέπει να εφαρμόσουν τους κανόνες που διέχουν τα ταμεία και πολλά, πολλές από αυτές τις πράξεις είναι δεσμευτικές και για τους ελεγκτές, κάτι που ε, προκαλεί αρκετή δυσαρέσκεια. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε οι βασικές πράξεις ε, να περιέχουν αρκετά στοιχεία ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Άλλο στοιχείο είναι το χρονοδιάγραμμα που ανέφερα νωρίτερα. Θα πρέπει να φροντίσετε οι κανονισμοί να υιοθετούνται όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα. Εάν έχουμε νέα πολιτική συνοχή, διότι πολλά κράτη-μέλη αντιστέκονται σε αυτήν. Εάν ε, λοιπόν έχουμε νέα πολιτική συνοχή, θα πρέπει να φροντίσουμε να ξεκινήσει εγκαίρως. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε την ίδια κατάσταση με σήμερα. Και τέλο, όσον αφορά του μηχανισμού υποβολή εκθέσεων, είναι αλήθεια ότι η πολιτική συνοχή είναι η μόνη πολιτική σήμερα με τόσο ισχυρό ε, ρυθμιστικό πλαίσιο. Έχει γίνει τεράστια δουλειά από όλε τι αρχέ διαχείριση, ε, έχουν ε, εκπονηθεί οι έχει γίνει τεράστια δουλειά και από άλλε μονάδε από τα τοπικά γραφεία κλπ ώστε η πολιτική συνοχής να αποδείξει ότι έχει αυτά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί πόλης εκθέσεων που μάλλον είναι κάπως υπερβολικοί και ίσως να μπορούμε να τους απλοποιήσουμε ή να τους κάνουμε πιο ομοιογενείς ε, ανάμεσα στο ERDF και το ESF για παράδειγμα. Και για το θέμα αυτό ε, συμπεριλαμβάνονται πολύ συγκεκριμένε προτάσεις ε, στην εκθεσή μας. Και τέλος, και δεν είναι μόνο δική μου θέση. Νομίζω ότι όλα τα μέλη της ομάδας ε, συμφωνούν. Ε, κάποιες από τις προτάσεις μας έχουν συμπεριληφθεί στον Γενικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Omnibus, αλλά υπάρχουν πολλές μη νομοθετικές προτάσεις ε, που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πολύ εύκολα ήδη τώρα, αλλά είναι θέμα βούλησης. σε όλα τα επίπεδα του συστήματος, ε, το ευρωπαϊκό, περιφερειακό, εθνικό, τοπικό κλπ. Βασιζόμαστε λοιπόν στην καλή βούληση όλων, διότι νομίζω ότι είναι προς κοινό μας συμφέρον το να απλουστεύσουμε την πολιτική αυτή. Από τώρα, πριν τις ευρωεκλογές, πριν σταματήσουν τελείως οι πολίτες να υποβάλουν ε, αιτήσει για τη χρηματοδότηση αυτή λόγω του υπερβολικού διοικητικού άχθους. Να κλείσω λέγοντας ότι η επόμενη έκθεση θα αφορά το λογιστικό έλεγχο. Θα μπορέσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε πολύ πιο αναλυτικές συστάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ. Ε, είμαι στη διάθεσή σας ε, για να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες ή να σας στείλω γραπτό στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Φυσικά ευπρόσδεκτη να επανέλθετε και στο μέλλον στην Επιτροπή μας. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε ένα σχέδιο γνωμοδότηση από τον κύριο Μαριζέ. Συγκεκριμένα, το θέμα της γνωμοδότησης είναι η διαχείριση των αλληλευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Τον Νοέμβριο του 2015 η Επιτροπή ΠΕΧ ε, στείλε μια αντιπροσωπεία στα υπερπόντια εδάφη σε εξόχως απόκεντρες περιοχές. Αποφασίσαμε έπειτα να συντάξουμε μια ιδέα πρωτοβουλία σε έκθεση για τη διαχείριση των αλληλευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ένα βασικό ζήτημα για την οικονομική ανάπτυξη. Η Ρέτζη θα συντάξει γνωμοδότηση, συνέταξε ε, την γνωμοδότηση αυτή ο κύριο Σομαριζή. Και τώρα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με ε, την παρουσίαση του σχεδίου κειμένου για τις 29 Νοεμβρίου. Α, όχι. Λάθος τα είπα. Τέλος πάντων, Νοεμβρίου. Το Μάρτιο θα γίνει ψηφοφορία στην Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή. Κύριο έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, πράγματι. Είμαστε στο πλαίσιο μιας πρώτης ανταλλαγής απόψεων μετά από την απόφαση να εκπονηθεί έκθεση από την Επιτροπή Αλλιές για τη διαχείριση των αλληλευτικών στόχων σε εξόχους από κέντρες περιοχές και η δική μας η, Περιφερειακή Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδότηση. Όπως είπατε, η έκθεση θα συνταχθεί μετά από την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αλίας με πρόεδρο τη συνάδελφό μας, την Ουλρίκη Ρόντουστ. Έγινε στη Ρεουνιόν συγκεκριμένα τον Νοέμβριο η επίσκεψη αυτή και εκεί τα μέλη της Επιτροπής Αλίας ήμουν και εγώ μαζί. Λάβαμε την πρωτοβουλία μετά να προτείνουμε τη σύνταξη έκθεσης. Και αυτό είναι και το θέμα που μας απασχολεί σήμερα. Γιατί? Πολύ απλά διότι διαπιστώνεται πως οι αλίες εξόχως από κέντρες ε, περιοχές έχει μέλλον μπροστά της. Υπάρχουν όμως και προβλήματα, φραγμοί που φρενάρουν τη βελτιστοποίηση των πλονεκτημάτων των περιοχών αυτών. Εξού και το διακύβευμα. Να μπορέσουμε να επεπιδίσουμε αυτά τα εμπόδια, στους φραγμούς, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερο να βελτιωθεί η νομοθεσία και η ρύθμιση. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε την πλήρη διάσταση των εκτιμάτων αυτών των περιοχών. Συνολικά, ισπανικά, γαλλικά, πορτογαλικά υπερπόντα διαμερίσματα είναι για την Ένωση μια έκταση πάνω από 2,7 εκατομμύρια χιλιόμετρα γονικά. Και φυσικά είναι πολύ σημαντική αυτή η περιοχή. Είναι και πάρα πολύ σημαντικά τα αλλιευτικά τους, οι τους δυνατότητες. Είναι σημαντικός ο αλλιευτικός τόλος. Ωστόσο, Η ελευτική στόλη των ξόχων από περιοχών είναι από τους λιγότερο ανεπτυγμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η μικρή παράκτεια κλίμακα σαλία είναι το 97% των ε, σκαφών στις εξόχους από κεντρές περιφέρειες. Ενώ στον Ατλαντικό είναι το 51% γιατί υπάρχει ένα περιθώριο ε, πρόοδου πολύ σημαντικό. Στη Ρεουνιόν συνολικά για το 2012 τα αποθέματα, μάλλον τα αλλιεύματα ήταν 0,5% το πολύ, επαναλαμβάνω 0,5% των αλλιευμάτων ε, στον Ινδικό ωκεανό για το ίδιο έτος. Και οι υπόλοιπες, τα υπόλοιπα αλλιεύματα ε, είναι από είτε ξένους είτε ευρωπαϊκούς στόλους. Άρα η κατάσταση ε, στις από απόκεντρες περιοχές είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς όμως, ακόμα πιο πολύ, ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο πρέπει να διερωτηθούμε ποια είναι η απόδοση των επενδύσεων που εδώ και χρόνια γίνονται σε αυτές τις από απόκεντρες περιοχές. Όταν βλέπουμε αυτή την πολύ τραγική θα τη χαρακτήριζα ε, κατάσταση. Είχαμε ανταλλαγές απόψεων με τον Επίτροπο Βέλα, την Επίτροπο Κρέτσου και τον Πρόεδρο Γιούγκερ. Και τους είπα Αυτή είναι η τελευταία η έσχατη ευκαιρία να κάνουμε κάτι, να μπορέσουμε να ε, βελτιώσουμε τους κανονισμούς κατά τρόπον ώστε οι επενδύσεις να συνδράμουν στην εξέλιξη, στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Βέβαια, δεν θα κάνω στη δική μου γνωμοδότηση τη δουλειά της Επιτροπής Αλίας. Δεν είναι αυτή η δική μας ε, δουλειά. Στην Επιτροπή Ρέτζι, έχουμε να πούμε πολλά σε σχέση με τους κανόνες, για τα είδη κτλ. Απλά θα πρέπει να προσέξουμε πολύ με τη δική μας γνωμοδότηση να εστιάσουμε στα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης. Συνεργάζομαι με εξαιρετικό τρόπο με τη συναλφολούρη και έτσι ώστε οι διαφορετικές εκθέσεις να είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Επιτροπή μας, νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουμε αυτό που έχω ήδη ξεκινήσει να κάνω εγώ, δηλαδή πώς αντιμετωπίζετε το ζήτημα της ε, τα επιχειρησιακά προγράμματα. Και οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να ενισχύσουν τις επενδύσεις για τις υποδομές, έτσι ώστε πραγματικά να διατηρηθεί ο κλάδος και να βοηθήσουμε ε, να προωθηθεί μεταποίηση των ψαριών επιτόπου, η διάθεση στο εμπόριο δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι ανήκωστα αυτά που γίνονται εκεί, στις έξω από κεντρές περιοχές. Να εισάγονται ψάρια, ενώ βρίθουν ψαριών τα νερά των περιοχών εκεί. Και μάλιστα τα ψάρια εισάγονται από πολύ μακρινές χώρες επειδή δεν υπάρχουν δομές για να μεταποιούνται επιτόπου τα προϊόντα αυτά και να δημιουργηθεί αυτός ο κλάδος που θα συνδέει αλίευση και ε, διάθεση του ψαριού στην τροφική αλυσίδα. Φυσικά και θα πρέπει οι τοπικές αρχές, περιφερειακές αρχές των διαφόρων κρατών μελών να ενισχύσουν τις επενδύσεις στις ε, λιμενικές υποδομές για τη μικρή κλίμακα παράκτη αλία. Εγώ βλέπω ότι εκατομμύρια ολόκληρα έχουν επενδυθεί σε κάποιες λεπτομέρειες ε, για τα εμπορευματοκιβώτια και κάποιες πύλες από που θα περνάνε στα λιμάνια. Αλλά τι κάνουμε για να βελτιώσουμε τα λευτικά σκάφη και τα λευτικά εργαλεία. Πρέπει λοιπόν να γίνει σωστή επιλογή. Διότι βλέπουμε ότι άλλα νησιά που έχουν τις κατάλληλες υποδομές ε, εποφελούνται Υπάρχει θέμα ρύθμισης και έχουμε και το άρθρο 349 της συνθήκης. Η Επιτροπή μας είναι αρμόδια για να εξετάσει όλα όσα άπτονται του άρθρου αυτού. Πώς έχει τώρα η τρέχουσα κατάσταση. Στις εξόχως απόκεντρες περιοχές απαγορεύεται η ανανέωση των λευτικών στόλων δυνάμει των κανόνων που ισχύουν σε ολόκληρη την νοσιακή επικράτη, δυνάμει της κοινής πολιτικής. Όμως, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ιδιαίτερη κατάσταση. Πολύ ξεχωριστή. 0,5 σας είπα σε των αλληλευμάτων από τους αλλείς μας. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν, αλλά να μην θέσουμε και υπό αμφισβήτηση τις βασικές αρχές της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να μην αποσυνδέσουμε τους στόχους περιβιωσιμότητας από τις άλλες μας προσπάθειες. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο μέσα θα πρέπει να βρούμε συμβαστικές λύσεις με βάση τη χρήση του άρθρου 349 για να θέσουμε όρους, προϋποθέσεις, αλλά παρόλα αυτά παράκτη αλική ε, και μικρής κλίμακας αλία να μπορέσει να ε, προβεί σε εξυγχρονισμό ανανέωση του στόλου. Αυτά είναι άκρος απαραίτητα πράγματα για τις εξόδους απόκεντρες περιοχές που πιστεύω ότι μπορούν να έχουν μέλλον. Πρέπει όμως να μπουν κάποια μέτρα και κάποιοι περιορισμοί. Γιατί έχουμε το 349 που δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια αποσύνδεση από τις βασικές αρχές των κοινοτικών πολιτικών σε όλους τους τομείς. Είτε στη γεωργία, είτε στην αλία. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία τα οποία θα ήθελα να συμπεριλάβω στην νομοδότησή μου και τα θέτω υπόψη των συναδέλφων για τη συζήτηση. Σας είπε η Πρόεδρος ποια είναι ε, η προθεσμία, ποιο είναι το πρόγραμμα. Ελπίζω όλοι μαζί οι συνάδελφοι να βοηθήσουν ώστε να έχουμε μια καλή γνωμοδότηση και είμαι στη διάθεσή σας ως συνήθως. Ευχαριστώ. Σκιώδης. Πόγκα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Θα ευχαριστήσω τον Γιουνούς για την δουλειά την οποία έχει κάνει και να του πω ότι ήξερα ότι θα συνεργαστώ μαζί του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη διαχείριση του ε, αλλιευτικού στόλου στις απότερες περιφέρειες. Είμαι πεπισμένος ότι ο τομέας της αλίας μπορεί να συνεισφέρει στην αηφόρο ανάπτυξη των απότερων περιφερειών. Γι' αυτό είναι απαραίτητο οι αλλοί μας να βοηθούνται γιατί ακριβώς τα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών απαιτούν μέτρα ειδικά όπως το είπε ο Μερζή, προβλέπει και το 349 της συνθήκης. Πριν τελειώσω θα ήθελα να σας πω ότι έχω τη χαρά να οργανώνω σήμερα μια συνάντηση η οποία θα επιτρέψει σε εκπροσώπους των αλλιέων από τις απότερες περιοχές να παρουσιάσουν τα ειδικά τους χαρακτηριστικά. Στις 12.30 θα ξεκινήσει η συνάντηση στο 6Q1, 6Q1. Σας προσκαλώ λοιπόν αγαπητοί φίλοι να έρθετε εκεί για να μπορέσετε να δείτε και ποιες είναι οι προκλήσεις της αλληλείας στις περιφέρειές μας. Thank you. Thank you for this kind invitation. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενή σας πρόσκληση και θα προχωρήσουμε στους κοιόδης εισηγητές. Ε, η κυρία Μπρέσο, παρακαλώ. Είμαι η σκιά της σκιάς. Very Yes, very visible. Merci, Madame la Présidente. Je vais... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του κ. Μασκούρα, ο οποίος μου ζήτησε να τον αντιπροσωπεύσω, μου άφησε ένα κείμενο το οποίο θα στείλω στον εισηγητή Τον ευχαριστώ λοιπόν και εγώ και ο Σκιώδης για τις εξαιρετικές του προτάσεις. Είναι οι κατάλληλες για την Επιτροπή μας, η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη της υπαίθρου και παρουσιάζει τις θέσεις μας με σωστό τρόπο. Εξ ονόματος λοιπόν του Σκιώδους Ξέρετε ότι και εγώ ασχολούμαι με τις απότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι περιφέρειες αυτές και γι' αυτό θα υπογραμμίσω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπογραμμίσουμε τη σημασία της αλίας για μια ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στις περιοχές αυτές. Και ο Σκιώδης τονίζει ότι η ανάπτυξη της αλίας στις περιοχές αυτές είναι κάτι το κρίσιμο γιατί δημιουργεί και θέσεις εργασίας αλλά επιτρέπει μια ανάπτυξη της υπαίθρου χώρας με αηφόρο τρόπο. Δεν μιλάμε για μεγάλους αλλιευτικούς τόλους. Μιλάμε για παραδοσιακές μορφές αλλίας, σημαντικές όμως για την ανάπτυξη της υπαίθρου περιοχές αυτές ο κ. Μάσκο σημειώνει ότι σε αυτές τις απότερες περιφέρειες λέγουμε ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στις αγορές, ενώ σε αυτή την περίπτωση η λογική είναι εντελώς διαφορετική. Οι ευκαιρίες υπάρχουν, οι θαλάσσιες ζώνες γύρω από τις περιφέρειες αυτές είναι σημαντικές, και το δυναμικό τοπικής ανάπτυξης είναι δεδομένο και γι' αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί σαν κάτι το πολύ σημαντικό για την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με αυτά που προβλέπει το 349. Βασικός στόχος της έκθεσής σας είναι ακριβώς αυτός να είμαστε σίγουροι ότι το δυναμικό αυτό μπορεί να γίνει πραγματική ανάπτυξη. Να μην μείνουμε σε θεωρητικό επίπεδο. Υπάρχουν περιφέρειες όπου τα πράγματα πάνε καλύτερα όπως τα Κανάρια, υπάρχουν άλλες περιφέρειες όπου τα πράγματα δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως. Αυτό που θα ήταν άσχημο για αυτές τις περιφέρειες Είναι λοιπόν να συνεχιστεί η ανάπτυξη του δυναμικού αυτού. Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε με συγκεκριμένο πια τρόπο να ξεπεράσουμε τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα bien sûr, de, de ce secteur de, euh, des fisheries, des, des mm, secteur de la pêche euh, dans les zones. Έτσι θα αναπτυχθεί η αλληλεία στις απότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Θα σας στείλω και το σημείωμα της ε, σκιώδους, του σκιώδου συγητή, αλλά θα τα συζητήσετε και στη συνάντηση. Ο επόμενος ομιλητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του πάνω σε αυτήν την γνωμοδότηση ε, που νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερη στο πλαίσιο της Ρέτζη, ε, αλλά ε, μεγάλο ενδιαφέρον για όσους συμμετέχουν άμεσα. Η ECR ε, καταλαβαίνει ότι οι ελευτικοί στόλοι στις εξόχους αποκτές περιοχές υπέφεραν από έλλειψη επενδύσεων στο παρελθόν, ε, τη δεκαετία του 70 και του 80 ε, και λόγω της, των περιορισμών της κοινή αλληλευτικής πολιτικής κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 90. Γι' αυτό επικροτούμε τις προσπάθειες να εξετάσουμε τις ρυθμίσει και θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή ώστε στην, στη γνωμοδότηση αυτή να διαπιστώσουμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω διατηρώντας ε, το, τα όρια του προϋπολογισμού. Επίσης, ε, το ECR ενδιαφέρεται να δει πώς ε, οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να βοηθήσουν στην εξέβρεση λύσης. Η προσέγγιση αυτή είναι νέα, αλλά έχουμε δει ότι έχουμε δει θετικέ ε, αλλαγέ σε διάφορα μέρη με την προσέγγιση αυτή. Πιστεύουμε ότι απομένουν και άλλα να γίνουν, ώστε οι άνθρωποι σε τοπικό επίπεδο να είναι οι κύριοι παράγοντε. Ε, αυτό αναφέρθηκε και κατά το EuroCities. Ε, όσον αφορά την περιφερειακή χρηματοδότηση, σε τοπικό επίπεδο γνωρίζουν καλύτερα οι άνθρωποι ποιε είναι οι ανάγκε και θα πρέπει η ενδυνάμωση των ανθρώπων σε αποκέντρες περιοχέ να αποτελεί προτεραιότητα της ε, ε, έκθεσης. Ε, Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να αναφέρω και κάποιες ε, διαφωνίε και αντιρρήσεις ε, του ECR για να προσπαθήσουμε να βρούμε συμβιβασμό σε διάφορους τομείς. Έχουμε αντίρρηση εδώ και πολύ καιρό όσον αφορά την ε, ειδική μεταχείριση των ιδιαίτερα αποκεντρών περιοχών που αναφέρεται στο άρθρο 49, διότι πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσουν σε στοχευμένα μέτρα που να λαμβάνουν υπόψη τις ε, ιδιαίτερες ε, συνθήκες ε, στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Έχουμε όμως κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά το άρθρο 394, διότι πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν περιφερειακές που δεν έχουν αυτά τα πλεονεκτήματα. Δεν έχουν το ίδιο όνομα και γι' αυτό θεωρείται ότι δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο, ο, ο ορισμός των ιδιαίτερα απόμακρων περιοχών είναι, ε, είναι αυθαίρετος. Η ομάδα ECR λοιπόν δεν είναι υπέρ μιας γνωμοδότησης REG ε, που προβλέπει την ε, περαιτέρω χρήση του άρθρου 394. Επίσης ε, η ομάδα μου έχει αντιρρήσει όσον αφορά ε, ένα νέο πρόγραμμα POSI ε, που να επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην αλληλεία ή την ανανέωση του στόλου στις ε, εξόχους από κέντρες περιοχές θεωρούμε ότι μπορεί να δημιουργήσει απλά άλλο ένα επίπεδο γραφειοκρατίας ε, αντί να προσφέρει από τα αποτελέσματα. Επίσης πιστεύουμε ότι λαμβάνοντα υπόψη τον περιορισμένο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τις ε, πληρωμές των επομένων ετών, ο συνολικός αντίκτυπος τέτοιων προγραμμάτων φαίνεται να μην εκτιμάται αρκετά. Πάντω, Γιούνου, σε ευχαριστούμε και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία μαζί σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω τους άλλους και όδης ε, εισήγητες. Άρα να δώσω τώρα στην κυρία Κρέλ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν ξέρω πολλά πράγματα για την αλληλεία, αλλά έχω μία ερώτηση προς τον ε, συντάκτη. Είπατε κατά την εισαγωγή σας ότι οι εξόχως απόκεντρες ε, περιοχές ε, έχουν πολλά ψάριες περιοχές τους, αλλά τελευταία φορά που βρέθηκα στις ε, Αζόρες, οι Αλίες παραπονούνταν ότι η μεγάλη στόλη της Ισπανίας κλπ. Ε, έχουν αδειάσει από ψάρια τα ε, διεθνή ύδατα, ε, δεν αλλιεύουν με βιώσιμο τρόπο και ότι αυτό είχε σημαντικές επιπτώσεις στις δικές τους ακτές. Αυτό είναι αλήθεια και εάν ναι, τότε ίσως θα πρέπει στη γνωμοδότησή σας να αναφέρουμε ότι για την περιφερειακή ανάπτυξη είναι απαραίτητη η βιώσιμη αλληλεία και στην Επιτροπή Αλληλείας να πούμε ότι δεν μπορούμε να προωθήσουμε την αλληλεία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές αν δεν υπάρχουν ψάρια εκεί. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό όντως ισχύει. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω εκπροσώπηση της ταμάρε. Εσείς παρακαλώ. δεν είναι ακόμη εδώ. Έρχεται ο εκπρόσωπος της Γαμαδέλτα Μάρε. Λοιπόν, με κρίμα. Τι να κάνουμε, λέει ο πρόεδρος. Θα λάβουμε μέρος στη συζήτηση όταν έχουμε την έκθεση του εισηγητή πλέον στα χέρια μας. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ομαγζέ. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για τις παρατηρήσεις σας. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα τα σχόλια. Μέχρι το 1990 αυτές οι ακροσαποκέντρες περιοχές δεν είχαν λάβει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με επενδύσεις για τον αναλυτικό στόλο τους, μόλις από τότε και μετά, το 1990, έγιναν δικαιούχοι και αυτές οι περιοχές. Έκτοτε λοιπόν παίρνουν αυτά τα κονδύλια. Όμως τότε ξεκίνησε ταυτόχρονα να λαμβάνονται, ξεκίνησαν να λαμβάνονται μέτρα πολύ έντονα σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα. Και επομένως ε, την πλήρωσαν διπλά κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα οι περιοχές αυτές. Το είπα και το ξαναείπα και επιμένω Φυσικά και δεν θέλουμε να μην ε, ισχύουν οι κανόνες βιωσιμότητας για τις περιοχές αυτές. Σε καμία περίπτωση είναι αυτός ο στόχος. Απλά θέλουμε να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος και ιδίω το δυναμικό αυτό, στο βαθμό του δυνατού, να μπορέσει να συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην τοπική ανάπτυξη. Πολλά και ενδιαφέροντα ακούστηκαν, Ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάγκη να πλουστευθεί ο κανονισμός. Βλέπουμε πολύ καλά ότι μόνο όταν μπορέσουμε να παγιώσουμε, να δρεώσουμε κλάδους ε, έχουμε ανάπτυξη. Όμως υπάρχει μεγάλη πολυπλοκότητα σε επίπεδο κανονιστικό και πολύ έντονοι περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτού του κανονισμού. Και αυτό πολύ συχνά οδηγεί σε απομόνωση του αλής, αφού άλλοι κλάδοι ε, μετεγκαθίστανται και δεν μπορούν έτσι να τηρηθούν και οι στόχοι για την τοπική ανάπτυξη. Το ECR ξέρω τι πιστεύει για το άρθρο 349, δεν είναι κάτι καινούριο, το ξέραμε και το έχουμε ξανακούσει. Όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι άκρως από κέντρες περιοχές κατά κάποιο τρόπο είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι οι πρώτες που ε, και οι πιο ιδιόρυθμες τα έλεγα, δεν μπορούν να δοθούν ομοιόμορφες λύσεις. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις επιδόσεις. Ό,τι αφορά την αλία, κατάσταση στο Νοτιμισφαίριο δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση στο βόρειο ημισφαίριο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ισχύσει όλη η νομοθεσία, να ισχύσουν όλοι οι κανόνες. Και στο νότιο ημισφαιρινό, οι κανόνες αυτοί σχεδιάστηκαν και καθορίστηκαν κυρίως για το βόρειο ή καταρχάς για το βόρειο ημισφαίριο. Όταν ανακαλύφθηκαν αυτοί οι κανόνες ήταν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στη Μεσόγειο, στον Ατλαντικό, κτλ. Σήμερα οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται και στον Ινδικό ωκεανό και στον Ειρηνικό ωκεανό και στην Καραϊβική και πρέπει ενίοτε να αναγνωρίσουμε με απαράλογο τρόπο εφαρμόζονται. Γι' αυτό το άρθρο 349 είναι χρήσιμο. Διότι θα μπορούσε να επιτρέψει όταν έχουμε να κάνουμε το παράλογο των κανονισμών, θα μπορούσε να επιτρέψει σε αυτών των παραλογισμών. Ξέρουμε πώς αντιλαμβάνεται το ECR, τους, Ευρωπαίους, τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Άρα, με την ίδια λογική πρέπει να στηρίξει το ECR, το άρθρο 349, γιατί αυτό θα μπορούσε να εμπνεύσει και άλλες καταστάσεις και το έχετε πει κι εσείς για τις ορεινές περιοχές, για παράδειγμα. Euh, la commission régie. Euh, euh, Constance Rennes l'a dit, elle n'est pas experte sur les questions pêche et je ne suis pas d'accord. Ούτε κι εγώ είμαι εμπειρογνώμων στα ζητήματα της αλίας. Ε, απλά νομίζω ότι οι κανόνες της κοινή αλληλευτικής πολιτικής οφείλουν να ισχύουν για το σύνολο του αλληλευτικού στόλου της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν ήρθε εκπρόσωπος της ΓΔ Μάρη, άρα θα με ελέγξει ο εκπρόσωπός της όταν δεν εφαρμόζουν οι Ευρωπαϊκοί Αλληλευτικοί Στόλοι τους κανόνες αυτούς, μπορούν να τους επιβληθούν κυρώσεις. Απλά θα ήθελα γάμα τα Μάρια να το επιβεβαιώσει. Ισχύει όμως ότι σε ορισμένες ακρος ε, απόκεντρες ε, περιοχές διαπιστώνουμε ότι κάποιο μέρος ε, του στόλου δεν σέβεται τους κανόνες. Και έχετε και ένα άλλο πρόβλημα που είναι σημαντικό και αφορά την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μας απασχολεί μάλλον. Πρόκειται σε ελευτικές συμφωνίες που συνάπτουμε με άλλες χώρες και δι χώρες ΑΚΕ. Και εδώ, κατά κάποιο τρόπο, στρέφουμε τα νότα μας στις άκρος απόκεντρε περιοχές. Η συνεκτικότητα λοιπόν, συνέπεια των πολιτικών. Είναι κάτι, πολύ σημαντικό αν θέλουμε οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται στις ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές να είναι οι βέλτιστες δυνατές. Δεν ζητούμε παραπάνω χρηματοδότηση. Δεν το άκουσα να το πει κανείς από τις εξόχως κεντρικές περιοχές Ούτε οι αρχές ούτε άλλοι φορείς το έχουν ποτέ ζητήσει αυτό. Αυτό που θέλουμε, που θέλουν, είναι να έρθουν οι ρυθμιστικοί, διοικητικοί, νομικοί φραγμοί που εμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη της αλίας. Για να ολοκληρώσω, ο πολύ γνωστός σε όλους μας Ραϊμό Μπαρ μας έλεγε μην ξεχνάτε ποτέ ότι καταγεστε από νησιά που περιβρέχονται από θάλασσα, από νερό. Ναι, ισχύει αυτό. Όμως παραγνωρίζονται οι τεράστιες δυνατότητες της θάλασσας. Η θάλασσα και η αλία πρέπει να είναι ο βασικός πυλώνας της ανάπτυξης, ε, ιδίως της περιφερειακής ανάπτυξης, για τις χώρες αυτές. Όμως εδώ μιλάμε για περιφέρειες που έχουν ποσοστά ανεργίας ρεκόρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 60% των νέων στη Ρεουνιόν, μιλάμε για κάτω τους 25, χρόνων, των 25 ετών, που είναι άνεργοι. Μαρτινίκα, Γουαδελούπη, αντίστοιχα ποσοστά. Άρα είμαστε ένοχοι αν δεν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Τώρα, πώς θα την επιτύχουμε την ανάπτυξη, εντάξει, θα το δούμε, είναι άλλο θέμα. Τουλάχιστον όμω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ας δημιουργήσουμε τις πλέον συνθήκες. συνθήκε. από τη στιγμή που είναι σημαντική και η χρηματοοικονομική υποστήριξη. Ο στόχος λοιπόν είναι η απόδοση ε, και η απόδοση των κοινοτικών πολιτικών και η συνεπής άσκηση και εφαρμογή των πολιτικών αυτών. Η έκθεση της, της Ολυρή και είναι πεπισμένος ότι θα βοηθήσει να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσε η συζήτηση για το θέμα αυτό. Θα συνεχίσουμε τώρα. Όταν παρουσιάσετε την πρότασή σας, τότε θα αντιδράσει και η DG Μάρια. Τώρα η έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών που συναντήθηκαν χθε το απόγευμα. Οι αποφάσεις τους έχουν σταλεί χθε το απόγευμα Μπορούμε να εγκρίνουμε... Α, όχι, ο κύριος ρόι. Εγώ δεν έχω πάρει το... τα πρακτικά, αλλά από ό,τι θυμάμαι δύο σημεία. Πρώτον, για το Omnibus έγιναν κάποιες καλές συζητήσεις. στο σημείο 3 θα πρέπει να φαίνεται και το όνομα του συντάκτη. Να αναφέρουμε καλύτερα τον εισηγητή της Ρέτζη. Πρέπει να βάλουμε, εν πάση το έγγραφο με το όνομα του συντάκτη. Και δεύτερη παρατήρηση, η άποψη την οποία έχω εγώ σε σχέση με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στα πρακτικά λέτε ότι όλοι έχουν δικαίωμα να αντιδρούν πάνω σε αυτά τα θέματα και στην επόμενη συνάντηση θα τα συζητήσουμε εκ νέου. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει νόημα. Δεν υπήρξε συμφωνία πάνω σε αυτό. Είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες και ο καθένας μπορεί να σχολιάσει τις εκκρεμότητες αυτές. Αλλά μπορείτε όμως στην επόμενη συνάντηση της Ρέγκι να παρουσιάσετε το ψήφισμά σας, την πρόταση ψηφίσματος. Να ξεκινήσει και η διαδικασία για την κατάθεση τροπολογιών με αυτόν τον τρόπο. Αυτά. Ε, ελπίζω να έγινα αντιληπτός ε, έτσι ώστε να μην επιβραδύνουμε τις εργασίες μας. Και είναι πάντα δυνατό τον Φεβρουάριο να αλλάξει κανείς αν θέλει ας πούμε την ερώτηση και να προσαρμόσει την ερώτησή του. Εγώ έρχομαι εδώ από την ΕΚΟΝ, εκεί ψηφίσαμε ένα ψήφισμα και είπαμε μεταξύ των άλλων έχουμε την ψηφοφορία και για δύο ερωτήσεις. Μπορούμε να κρατήσουμε τη διαδικασία δηλαδή ισορροπημένη και δημοκρατική και να μην περιμένουμε δύο μήνες για σχόλια. Δεν ξέρω τώρα οι συνάδελφοί μου τι πιστεύουν για αυτά. Δεν ξέρω αν... Κοιτάξτε, Έχουμε μια ώρα μπροστά μας τουλάχιστον. Ας δουλέψουμε, ας μείνουμε εδώ να δουλέψουμε. Τι να πεις. Λοιπόν, για την προφορική σας ερώτηση εννοείται όχι. Όχι. Δεν θα ασχοληθούμε με την προφορική σας ερώτηση σήμερα. Εσείς μας θέσατε στην ημερήσια διάταξη τα πρακτικά. Τα πρακτικά λέγουν ότι ο καθένας μπορεί να σχολιάσει το κείμενο αυτό, την επόμενη φορά θα αποφασίσουμε κτλ. Δεν είναι σωστό αυτό. Τι θα πει αυτό, τίποτα δεν θα πει. Καταρχάς, συμφωνώ μαζί σας και είπα χτες κατά τη διάρκεια των συντονιστών ότι δεχόμαστε τα τέσσερα αυτά σημεία στην επιστολή και ότι θα συμπεριλάβουμε και τις επιμέρους προτάσεις μας για, για τον ορισμό των εισηγητών εισηγητριών θα προσθέσουμε τα ονόματα στον κατάλογο. Αυτό το αποφασίσαμε. Και μου το επιβεβαιώνει και η γραμματεία. Αυτά. Από ό,τι κατανοώ, λέει η Πρόεδρος, η Γραμματεία εφαρμόζει το άρθρο 54. και εμείς προσπαθούμε να βρούμε τους δικούς μας τρόπους εφαρμογής του 54 συν και τα λοιπά. Οι συντονιστές πιστεύουν λοιπόν ότι το 54 συν σημαίνει ότι ε, έχουμε ένα εισηγητή και θα προσθεθεί στον κατάλογο των ομιλητών για την συγκεκριμένη έκθεση. Για το δεύτερο θέμα, σχετικά με την πρόταση προφορικής ερώτησης, αυτό το οποίο αποφασίσαμε χθες είναι να δεχτούμε ότι θα συνεχίσουμε την εργασία μας πάνω σε αυτό στη Ρέτζη, ότι η Ρέτζη θα αναλάβει πρωτοβουλία με βάση τον εκπροσ... τις προτάσεις των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έτσι ώστε να υπάρξει μια προφορική ερώτηση και πρόταση ψηφίσματος εξ ονόματος της Ρέτζη. Εσείς λέτε ότι είσαστε διαθέσιμος και θα περιμένουμε ε, έτσι ώστε να λάβετε ε, προτάσεις και τροπολογίες από όλους όσους συμμετέχουν στη Ρέτζη. Αυτό δεν είπατε. Όλα αυτά που είπατε είναι σωστά. Αλλά εγώ είπα κι άλλα. Μας ζητείτε να κάνουμε μία πρόταση ψηφίσματος. έτσι ώστε να κάνουμε ένα κείμενο και να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, γιατί αλλιώς θα χάσουμε ένα-δύο μήνες. Έχω τέσσερις συντονιστές εδώ. Αν συμφωνούν οι άλλοι συνάδελφοι, θα τροπολογήσουμε τα πρακτικά λοιπόν, ότι θα εργαστούμε πάνω στις προφορικές ερωτήσεις, ότι οι τροπολογίες θα ληφθούν υπόψη και θα συνεχίσουμε την προετοιμασία του ψηφίσματος. Αυτό θέλετε. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Θέλω όμως να μου δώσετε και κάποιον από τη γραμματεία να με βοηθήσει. Φυσικά κύριε Βανίστελρόι. Ευχαριστώ λοιπόν. Με τις διορθώσεις αυτές... Ναι, κυρίες και κύριοι, λοιπόν διορθώνει η πρόεδρος. Με τις διορθώσεις αυτές λοιπόν διορθώνουμε τα πρακτικά. Έχετε κάτι στα διάφορα. Δεν έχετε τίποτα. Απίστευτο. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η επόμενη συνάντησή μας είναι η 3η 29η Νοεμβρίου, πρωί και απόγευμα. Να ευχαριστήσω την επιμελητία. Οι ψηφοφορίες θα γίνουν το απόγευμα στις 29 Νοεμβρίου. The votes will be at 3. I close the meeting. Thank you.